Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να σας παρακαλέσω να καθίσετε. And again, may I ask you to... Να σας παρακαλέσω να πάρετε τις θέσεις σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ρέγγι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σήμερα έχουμε μεικτή συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων από τα κράτη-μέλη. Επιτρέψτε μου να τηρήσω παρόλα αυτά την κανονική διαδικασία. Ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της, σημερινής της διάταξης της σημερινής συνεδρίασης και έχω μια ερώτηση για τα μέλη της Επιτροπής Ρέγγι. Έχετε κάποια πρόταση, ε, κύριε Βανίστελ Ρόι, από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά είναι να επιταχύνουμε λίγο για να περάσουμε στα πραγματικά στα θέματα. Να κάνω μια παρατήρηση για την περασμένη φορά ε, που να κάνω μια αναφορά στην περασμένη φορά που συζητήσαμε ε, τις καταστροφές της Αντίλες στο ε, Σεντ Μάρτιν και τώρα έχουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και το ερώτημα είναι πότε θα το συζητήσουμε. Είχα και το αίτημα από την κυρία Σπυράκη, ενδεχομένως θα μπορούσε να πει δύο λόγια γι' αυτό και να δώσουμε μετά χρόνο για τη συζήτηση, να βρούμε χρόνο για αυτή τη συζήτηση. Κυρία Σπυράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βανίστερ Ρόι για το ερώτημα αυτό που αφορά τον ελληνικό λαό. Ε, κυρία Μιχαήλοβα, θα ήθελα να σας ζητήσω να εισάγετε αυτό το σημείο για την Ελλάδα αύριο και θα ήθελα να το συζητήσουμε και στην Ολομέλεια, να το συμπεριλάβουμε στην Ολομέλεια μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Να πω στους συναδέλφους μας, στην Επιτροπή Ρέτζη, ότι είναι σημαντικό να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τον ελληνικό λαό, ζητώντας από την Επιτροπή να εξαιρεθεί από την Εθνική Συμβολή σε έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό σε σχέση με αυτή την καταστροφή και να τροποποιήσουμε τον κανονισμό όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Τα υπόλοιπα αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βανίστα Λερό, κυρία Σπυράκη. Από λοιπόν σήμερα έχουμε δύο αντιπροσωπείες Βουλγαρίας και Ρουμανίας πριν τις ψηφοφορίες ε, θα τους ακούσουμε, ε, θα τους δώσουμε ξεχωριστό χρόνο για μια εισαγωγή ε, και, και θα βρούμε και χρόνο για να κάνουμε μια παρουσίαση, να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και κατά τις συνεδρίες των συντενιστών έχουμε ήδη συμπεριλάβει ε, στο ημερήσια διαταξή για τους συντονιστές συζήτηση για ένα πιθανό προφορικό ερώτημα για την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Μπορούμε να Εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη με αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λοιπόν, εγκρίνουμε τα πρακτικά συνεδριάσεων, τα σχέδια πρακτικών των συνεδριάσεων της 9 και 10ης ε, ε, Οκτωβρίου είναι διαθέσιμα online. Προτείνω ως συνήθως, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις... Δεν θα περάσω τώρα σε ανακοινώσει τη Προέδρου, θα περάσουμε στα θέματα που είναι να συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών για το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020, ευκαιρίες, προκλήσεις και επόμενα βήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω όλους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα στην διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών για να συζητήσουμε ένα σημαντικό θέμα. Το μέλλον της πολιτικής συνοχής και πώς θα διαμορφωθεί μετά από την τωρινή χρηματοδοτική περίοδο και ε, μετά από το τέλος της το 2020. Ήδη έχουμε συζητήσει το θέμα εδώ στην Επιτροπή μας πολλές φορές, ε, με διάφορες ευκαιρίες. Επίσης έχουμε εκπονήσει ένα ψήφισμα που ονομάζεται ε, «Θεμέλη λύθη για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής μετά το 2020» που βασίστηκε στη δική μας έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που εκπονήσαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Αναφέρει την αρχική θέση του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια το Μάιο φέτο. Αυτή τη στιγμή μελετάμε την πρόταση Omnibus όπω ονομάζεται που σχετίζεται με την ενδιάμεση αναθεώρηση τη τρέχουσα περίοδου και η κυρία Κρέλ που θα μιλήσει αργότερα σήμερα είναι η συγγετρία τη Ρέτζη για το αρχείο αυτό. Όπω γνωρίζουμε, η 7η έκθεση συνοχή δημοσιεύτηκε στην, ε, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών τον Οκτώβριο. Και ήδη έχουμε κάνει μια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας μαζί με την κυρία Κρέτσου, την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με την Επιτροπή Κότερ της Επιτροπής των Περιφερειών. Η Επιτροπή μας επίσης ε, θα εκπονήσει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για αυτό το σημαντικό έγγραφο. Το 2018 οι εργασίες ε, για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα ξεκινήσουν και αναμένουμε τις προτάσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το Μάιο, όπως μας έχουν ενημερώσει. Αύριο θα γίνει μια συνεδρίαση, μια ακρόαση με τον κύριο Έτιγκερ, τον ε, Επιτροπό που είναι αρμόδιος για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελκύει, ελπίζω ότι θα λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Θα ήθελα επίσης να ρίξουμε μια ματιά στις βέλτιστες πρακτικές όπως αναδύονται από την τωρινή και τις προηγούμενες προγραμματικές περίοδου. Εμείς λοιπόν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσδοκούμε μια επικοδομητική όμορφη συζήτηση σήμερα και σας εύχομαι να έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις ε, σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε με τους ομιλητές, έχω κάποιες τεχνικές ανακοινώσεις για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, παρακαλώ συμπληρώστε το έγγραφο χρόνο Δώστε το στους κλητήρες. Τα έγγραφα αυτά θα τα βρείτε ε, μπροστά στα έδρανά σας. Είναι σαφές. τα δικά μας μέλη σας ξέρω ήδη. Είναι ευκολότερο να δω ποιος θέλει το λόγο. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Επίσης, όπως συνήθως, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία όπου οι συντονιστέ των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου θα λάβουν το λόγο, μετά τα μέλη του Εθνικού, των Εθνικών Κοινοβουλίων και μετά τα υπόλοιπα μέλη. Θα ήθελα να Καλωσορίσω τώρα θερμά την Επίτροπο κυρία Κρέτσου που είναι προσκεκλημένη μας σήμερα και θα συμμετέχει στη συζήτηση και θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω και να καλωσορίσω τον Υπουργό ΑΜΠ Υπουργό Αρμόδιο ε, Περιπολιτικής Συνοχής ε, της Εσθονικής Προεδρίας. Καλός φίλος της Επιτροπής Ρέτζη έχει ξανάρθει εδώ για να συζητήσουμε τα προβλήματα της πολιτικής συνοχής. μεγάλη μας ευχαρίστηση να μην σπαταλάμε άλλο το χρόνο. Το χρόνο μας σας δώσουμε το λόγο στην κυρία Κρέτσου για να μας κάνει κάποια σχόλια για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ το Ευρωκοινοβούλιο καθώς ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στη σημερινή συνεδρία. Σας ξέρετε πολύ καλά ότι για μας, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εθνικά κοινοβούλια δραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, στον δημοκρατικό έλεγχο των πολιτικών μας και τη μεταφορά τους ε, προς τους πολίτες μας. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπου και να πάω προσπαθώ να συναντηθώ με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, να εξηγήσω τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να διατηρήσω συνεχή και διαφανή διάλογο. Σήμερα συναντιόμαστε στο ναό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για ένα πολιτικό διάλογο. Κέρια σημασία είναι και η χρονική συγκυρία για την πολιτική μας, καθώς εδώ έχουμε έρθει για να συζητήσουμε για το μέλλον της πολιτική συνοχή μετά το 2020. Έχουμε λάβει ε, γνωμοδοτήσει από όλα τα κράτη-μέλη σχεδόν σχετικά με το μέλλον τη ε, πολιτική αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τη δουλειά που έχετε κάνει και την οποία εκτιμώ. Ιδιαίτερα εκτιμώ και το έργο της Επιτροπής ε, Ρέτζη, κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά εργάζεστε άοκνα και για την έκθεση Festival. Χρειάστηκε πολλή δουλειά, καθώς και γνωμοδότηση του κύριου Σνάιντερ. Μας έδωσε πραγματικά τροφή για σκέψη. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Κυρίες και κύριοι, Μπορούμε να δούμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μία, ε, έναν κόσμο με ειρήνη και ευημερία ανεφεργουμένο, όμως υπάρχουν γενικευμένες προκλήσεις, παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, οικονομικές και κλιματικές αλλαγές που έχουν δημιουργήσει εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αυξηθεί ε, οι ανισότητες, όπως βλέπουμε και στην τελευταία πλέον πρόσφατη έκθεση. Και όλα αυτά μπορεί να υποσκάψουν ε, τις βασικέ αρχές ε, πάνω στι οποίε χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτώντα προ το μέλλον, η απάντηση είναι δύο λέξει Πολιτική συνοχή, Γιατί είναι η πλέον απτή και ορατή έκφραση τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύης διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες σε όλες τις περιφέρειες. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε την τελευταίο μήνα την 7η έκθεση για την ε, κατάσταση σχετικά με τη συνοχή στην Ευρώπη και αναδεικνύονται τα εξή στοιχεία. Πρώτον, η σύγκληση ε, υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ αποσχόμενο για το μέλλον. Σημαίνει ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα την πολιτική συνοχή. Όμω, όλο παραδόξω, η έκθεση μα λέει ότι αυξάνονται οι ανισότητε μεταξύ χωρών και στο εσωτερικό των χωρών μεταξύ αστικών, και, αστικών περιοχών και της υπαίθρου μεταξύ μικρών πόλεων και των μεγαλοπόλεων. Αυτό είναι και ο λόγος που θεωρώ ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει ε, να συνεχιστεί ε, και να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε όλες τις περιφέρειες. Ξέρουμε ότι και η Επιτροπή Ρέτζη και πολλά κράτη-μέλη συμμερίζονται την ίδια γνώμη. Η έκθεση επίσης μας λέει ότι οι μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης ε, ενισχύονται. Κοινωνική συμπερίληψη, ένταξη των μεταναστών, κλιματική αλλαγή και ενέργεια, ε, βιώσιμες μεταφορές, βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, ψηφιακές υποδομές, καινοτομία και έρευνα. Αυτοί είναι τομείς στους οποίους η πολιτική συνοχή έχει κάνει τη διαφορά και θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον θα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε κράτη-μέλη και περιφέρειες να αυξάνουν την ε, ανθεκτικότητά τους και να προσαρμοστούν καλύτερα στις νέες τάσεις της οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης. Κυρίε και κύριοι, τώρα το θέμα είναι ε, πώς θα το κάνουμε αυτό. Πώς μπορούμε να επικεντρωθούμε σε απτά αποτελέσματα για να αφήσουμε ε, κατά μέρο ε, τους κανόνες και άλλες συνταγές. Πώς η πολιτική συνοχή θα γίνει απλούστερη για τους δικαιούχους, πιο ευέλικτη και έτσι φιλική προς τον δικαιούχο ποια είναι η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της αλλαγής και της σταθερότητας. Βλέπω ότι όλα ξεκινούν με την εμπιστοσύνη, που είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Εγώ είμαι υπέρ της ριζικής απλούστευσης της πολιτικής που δεν έχει αλλάξει εδώ και 25 χρόνια που κάποιες φορές ε, είναι φιάλτης για τους δικαιούχους. Πρέπει λοιπόν να απλουστεύσουμε τη διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου. Νομίζω ότι αυτό θα βρει το πρώτο βήμα για την ε, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ ε, αρχών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Για, το, για την πραγματική περίοδο 2014-2020 η προσέγγιση μας έχει δώσει υψηλά επίπεδα διασφάλισης, όμως βλέπουμε ότι είναι μακροσκελής και ε, επαχθείς διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν να τα αναθεωρήσουμε. Ε, το κόστος δεν πρέπει να είναι το, μοναδικό κριτήριο. Πολλοί στηρίζουν ένα σύστημα που ε, η Επιτροπή θα πληρώνει βάσει προσυμφωνημένων ε, όρων. Πρόσφατα είδαμε ότι οποιαδήποτε περιφέρεια μπορεί να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις παρότι υπάρχουν ε, κριτήρια τα οποία καθορίζονται στην αρχή τη πραγματική περίοδου, παίρνει πολύ καιρό να κάνουμε τις προσαρμογές και είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου ε, θα έπρεπε να έχουμε ανταποκριθεί πολύ πιο γρήγορα. Για παράδειγμα στη Βαλονία με την Caterpillar. Χιλιάδες εργαζόμενοι έμειναν χωρί δουλειά από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε φυσικέ καταστροφέ και άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται ευελιξία στο μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, μη διαθέσιμα ποσά ε, στο πλαίσιο της, επιτροπής, ε, της πολιτικής συνοχής μπορούν να καλύψουν ε, τρύπες. Η ευελιξία αυξάνεται και με ένα απλό κανονιστικό πακέτο όπου οι εφαρμοστέ κανόνε για τα διευθυντικά ταμεία είναι οι ίδιοι. Τέλο, θα ήθελα να επισημάνω το θέμα τη διακυβέρνηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι το, η χαμηλή ποιότητα διακυβέρνηση παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη ε, και μειώνει τον ε, αντίκτυπο τη ε, δημόσια επένδυση. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέω ότι δεν είναι το παν τα χρήματα πρέπει να επενδύσουμε και στη διοικητική μα ικανότητα. Γι' αυτό απευθυνόμαστε και στου εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί έχετε βαθιά γνώση των όσων συμβαίνουν ε, στι χώρε σα και τι εκλογικέ σα περιφέρειες, που είναι πολύτιμοι. Έχετε μέσα ε, τεχνογνωσία για την μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό πλαίσιο και έχετε έναν αποφασιστικό ρόλο για δραματίστε σε ό,τι αφορά ε, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. και είστε στην καλύτερη δυνατή θέση για να μας βοηθήσετε και εμά να βρούμε τα κατάλληλα κίνητρα για την υλοποίηση των ιδρυτικών μεταρρυθμίσεων. Κλείνοντα κύριε και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι να εργαζόμαστε από κοινού. Και αυτό το πρώτο βήμα είναι κάθε Ευρωπαίος πολίτης στις εκλογικές σας περιφέρειες να γνωρίζει ότι η πολιτική συνοχή ε, επιτυχάνει αποτελέσματα. Οι κοινέ ε, δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχουμε προτείνει με την Επίτροπο Τάισεν ε, φέρνουν αποτελέσματα στις περιφέρειες. Το σημαντικό τώρα είναι να παραμείνουμε αφοσιωμένοι και προσυλλομένοι σε αυτό το έργο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Εγώ δεν λέω να πλέξετε το εγκόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς ε, να αναφέρω την κατάσταση όσο έχει, και να λέτε, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, να αναφέρετε αυτό. Γιατί εδώ και πολύ καιρό πάντα κατηγορούμε τις Βρυξέλλες για όλα τα άσχημα και για όλα τα καλά είναι οι κυβερνήσεις και οι δήμαρχοι που τα έχουν καταφέρει. Και στη χώρα μου το ίδιο βλέπω. Πρόσφατα έγινε ένα τεράστιο σοου με επενδύσει. Το 90% βέβαια χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. κανεί δεν το λέει αυτό όμω. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα που να έχει επίτροπο και να μην τον προσκαλεί σε τέτοιου είδους ε, εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν βήματα στην επικοινωνία. Μίλησα τηλεφωνικώ με τον Επίτροπο Μοέδα. Ήταν στο Μάτσεστερ, σε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε επενδύσει 150.000 ε, ευρώ και δεν υπάρχει καν αναφορά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν ρώτησε λοιπόν ο Επίτροπο από πού προήλθαν αυτά τα χρήματα, ε, είπαν από το Δήμαρχο. 150 εκατομμύρια ευρώ είχαμε δώσει. Πρέπει λοιπόν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Πρέπει λοιπόν να ξεκολουθούμε να εξηγούμε την πολιτική συνοχής. Οι συνάδελφοί μας από την Επιτροπή των Περιφερειών νομίζω με τα χαρά θα σας δώσουν ε, λεπτομέρειες για την ε, συμμαχία συνοχής ε, που έχω προτείνει στις αρχές της χρονιάς και είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται. Τέλος, να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος Γιούγκερ την περασμένη εβδομάδα θέσπισε μία task force για την επικουρικότητα και αναλογικότητα, όπω είχε ανακοινώσει στην ομιλία του για την κατάσταση τη Ένωση το Σεπτέμβρη, και θα παρτίζεται από μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτή η task force είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και απηχεί ε, τα βασικά μηνύματα του πολιτικού μας διαλόγου. Έτσι μπορούμε να δούμε πώς η πολιτική συνοχή θα είναι πιο σαφής, αποτελεσματική και με προσταθεμένη αξία. Ε, είμαι σίγουρη ότι η συζήτηση θα είναι ιδιαίτερα γόνιμη. Αυτή εδώ η Επιτροπή είναι μία από τις καλύτερες. Ε, με, ε, απαρτίζεται από οι δήμονες που δουλεύουν επί τόπου, ξέρουν τι πάει και τι δεν πάει καλά και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής, Εθνικών Κοινοβουλίων και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρέμβαση και τα σημαντικά μηνύματα που μας δώσατε. Αν δεν απατώμε, πρέπει να φύγετε σε λίγο. έχουμε να συζητήσουμε και τα θέματα της στρατικής των Άλπων, μάλιστα. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην δική μας την συνεδρίαση και από τη, τουλάχιστον έχω καταλάβει ο διευθυντή τη ΓΔΡΕΤΖΙ, ο κύριο Φονμπρέσκα, θα μείνει μέχρι τέλου. Άρα θα υπάρχει πρόσωπο τη Κομισιόν να απαντήσει σε ενδεχόμενα ερωτήματα. Ο κύριος Φονμπρέσκα είναι και από τους ομιλητές μας στη συνέχεια. Και τώρα έχω τη μεγάλη χαρά να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή μας, ε, τον κύριο Γιάκ Αμπ, Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, εκ μέρους ε, της Αστονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν την προσέγγιση της Προεδρίας του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο κύριε Αμπ. Κυρία Μιχαήλοβα, κυρία Επίτροπε, Κρέτσου, Αγαπητοί ευρωβουλευτέ και Εθνικοί βουλευτέ, πρώτα απ' όλα θέλω να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο σεμινάριο για το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Θέλω να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συζητήσω μαζί σα τι ευκαιρίε, τι προκλήσει και τα επόμενα βήματα. Και είναι και η κατάλληλη χρονική στιγμή για μια τέτοια συζήτηση, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντο ε, το προσεχέ πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει και την πολιτική συνοχή. Προτού έρθω όμως στην ουσία του ζητήματος, στο θέμα δηλαδή τη σημερινή ημερίδα, θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Μιχαήλοβα, την κυρία Κρέλ και όλου του κοιόδε εισηγητέ για μια εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου για το κανονισμό όμνibus. Πετύχαμε πολλά σε ό,τι αφορά την απλούστευση ε, του γενικού κανονισμού. Τον Ιούλιο Οπότε και παρουσιάσαμε τις προτεραιότητες της Αστωνικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ προσωπικά σας είχα πει ότι ένας από τους στόχους της Προεδρίας είναι η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής με επίκεντρο την απλούστευση της εφαρμογής πολιτικής συνοχής και πράγματι είναι ένας στόχος που πετύχαμε. Το θέμα το συζητήσαμε σε διάφορα επίπεδα και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα. συζητήσαμε εκεί κυρίως τα θέματα που άπτονται της πολιτικής συνοχής. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συνεδρίασε ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που μου δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να σας εκθέσω τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε σε, αυτό, σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε ένα έγγραφο συμπερασμάτων για τις συνέργειες ε, στην πολιτική συνέχιση μετά το 2020. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, πολιτικές ε, που πρέπει να αλληλοσυμπληρούνται. Πρέπει να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και μηχανισμών οι βασικοί κανόνες ε, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Είναι μια ιδέα και αυτό ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής των διαφόρων ταμείων μηχανισμών το ε, συστήνει και η ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση ώστε οι δικαιούχοι πιο εύκολα να μπορούν να, να βρουν το δρόμο τους σε αυτό το πολύπλοκο δύσβατο τοπίο της ε, χρηματοδότης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρμόδιοι για θέματα συνοχής ε, υπουργοί εξέτασαν την προηγούμενη εβδομάδα την 7η έκθεση συνοχής και τα ζητήματα που αφορούν και το προσεχές πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με τα μπορώ να σας πω ότι οι συζητήσει ήταν ειλικρινεί και ενδελεχεί. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν πως η πολιτική συνοχή έχει να διδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ε, μείωση των ε, ανισοτήτων και την προώθηση των διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων και της ανταγωνιστικότητας. Δεν πρέπει πάντως να επαναπαυόμεθα στις δάφνες μας. Πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να καλύψουμε τα κενά ε, που υπάρχουν στο μέτωπο της ανάπτυξης. Μετά την ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων μπορώ να σας πω ότι είναι αντιληπτή η σημασία της πολιτικής συνοχής και το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί ως προς τους κανόνες ε, που διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να τους καταστήσει πολύ πιο απλούς. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ώστε οι κανόνες να είναι απλοί, ευανάγνωστοι και να μην είναι δυσκίνητη, να είναι ευέλικτη σε σχέση με το προσεχέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποιε είναι τώρα οι προκλήσει και ποιε είναι οι ευκαιρίε. Με βάση την 7η έκθεση συνοχή, οι περιφέρειε, τα κράτη-μέλη, αλλά και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελούνται από την πολιτική συνοχή. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρώπη, όπως είπε και η Επίτροπος Κρέτσου, περιφέρειες που υπολείπονται σε οικονομική ανάπτυξη και όπου τα ποσοστά ανεργία είναι υψηλά. Επιπροσθέτω, υπάρχουν νέε προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη, να τονώσουμε την καινοτομία, να αυξήσουμε τα ποσοστά απασχόληση και να καταπολεμήσουμε ιδίω την ανεργία των νέων και βέβαια να μειώσουμε και τη φτώχεια. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι θα πρέπει να είναι αναλύωτη η απομονωμένη από την πραγματικότητα η πολιτική συνοχή. Το αντίθετο, το έχουμε αντιμετωπίσει με νέε προκλήσει. Άρα χρειαζόμαστε ολοκληρωμένε λύσει. Λύσει οι οποίε ε, θα περιλαμβάνουν διάφορου τομεί, διάφορα ταμεία και κονδύλια. Και η πολιτική συνοχή πρέπει να είναι και αυτή ευέλικτη, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στι πραγματικέ ανάγκε των περιφερειών και των κρατών. Εκτό τη ευελιξία, πρέπει να εγγυηθούμε και την πολιτική σταθερότητα, διότι η πολιτική συνοχή έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά και τι μακροπρόθεσμε επενδύσει και την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η πολιτική συνοχή προφανώ και δεν αποτελεί πανάκια για όλα τα προβλήματα. Πρέπει να είναι στοχευμένη. Πρέπει να έχει σαφεί στόχου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα για το τι πολιτική επιθυμούμε και για το ποια θα πρέπει να είναι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε θα είναι η προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων. Σαφή, ορατά αποτελέσματα που δημιουργούν μεγαλύτερη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και καταδεικνύουν στους πολίτες τι ωφέλη έχουν αποκομίσει ή θα αποκομίσουν και οι προσωπικά και οι περιφέρειές τους δύσκολο να υποτιμηθεί η σημασία και της διασυνοριακής συνεργασίας στην πολιτική συνοχή. Πάνω από το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε μεθοριακές περιοχές. Οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλο δυναμικό σε ό,τι αφορά την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. και ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και προσώπων. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξέβρεση λύσεων στα διασυνοριακά προβλήματα είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Αγαπητοί φίλοι, η πολιτική συνοχή αποδείχθηκε ότι συνιστά σημαντική προστέμενη αξία και αυτό βάσει και τη πολιετούς προσέγγιση, ε, τη συνεκτικότητάς τη με τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η πολιτική συνοχή ε, είναι από τους ε, πρωτοπόρους σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και σίγουρα η πρόοδος αυτή πρέπει να αναγνωριστεί αλλά και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερε συζητήσει γίνονται για το μέλλον τη πολιτική συνοχή και είμαι πεπισμένο πω από κοινού όλοι μαζί θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε κατά τέτοιον τρόπο την πολιτική συνοχή ώστε να βελτιώσει την ανάπτυξη των χωρών μας, των περιφερειών μας, άρα να βελτιώσει κατά συνέπεια και την ευημερία των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δώσετε να σας μιλήσω για τα θέματα που μας απασχόλησαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αμπ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε και για τα μηνύματα που δώσατε, να αποχαιρετήσουμε την Επίτροπο και να συνεχίσουμε με τις εργασίες μας. Um, now I, I uh, go to uh, the, the next part of our debate today. Ας περάσουμε στο επόμενο μέρος της ε, συζήτησής μας. Έχουμε πέντε πολύ ενδιαφέροντες ε, ομιλητές ε, που θα μας παρουσιάσουν τις διαφορετικές ε, προσεγγίσεις της πολιτικής συνοχής, βέλτιστες πρακτικές και οράματα για το μέλλον. Οι πέντε αυτοί οι ομιλητές είναι ο κύριος Έρικ Βον Πρέσκα, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή η Κομισιόν προετοιμάζει τις μελλοντικέ προτάσεις πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020. Η ομιλία του λοιπόν ε, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Και δεν βλέπουμε την ώρα να μάθουμε τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επόμενη ομιλήτρια θα είναι η κυρία Ιβελίνα Βασίλεβα, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ιδάτων στην Εθνοσυνέλευση της ε, Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Θα μας πει κάποια πράγματα για τις βουλγαρικές απόψεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, δίνοντας μας και κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Η κυρία Ροβάνα Πλάμπ είναι πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας. Η Ρουμανία θα έχει την Προεδρία την Άνοιξη του 2019. Μια περίοδο κλειδί για την προετοιμασία της επόμενης χρηματοδοτικής περίοδου. Η Βουλγαρία θα πάρει τη σκητάλη της Προεδρίας τον Ιανουάριο του 2018 και η Ρουμανία θα συνεχίσει το έργο στις αρχές του 2019. Ο κύριος Μίχαελ Σνάιντερ είναι μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, πολύ καλός φίλος της Επιτροπής μας εδώ στις Ρέτζες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η συγητής ε, της Επιτροπής των Περιφερειών για τη γνωμοδότηση που αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που θα ακούσουμε και τη φωνή της Επιτροπής των Περιφερειών εδώ. Τέλος, η κυρία Κωνσταντς Κρέιλ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας, συντονίστρια της πολιτικής της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης είναι η συγγήτρια για τα βασικότερα έγγραφα της Επιτροπής, το φάκελο Omnibus. Καλωσορίζω λοιπόν τους ομιλητές μας. Πρώτος ομιλητής ο κύριος Φομπρέσκα. Έχετε το λόγο κύριε Φομπρέσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Θα είμαι πολύ σύντομος και θα αποφύγω να επαναλάβω τα όσα μας είπε μόλις η Επιτροπός μου. Προτείνω λοιπόν να εστιαστώ σε τέσσερα σημεία τα οποία αφορούν ιδιαίτερα ε, την Κομισιόν ε, και την απασχολούν ε, καθώς προβληματίζεται για το μέλλον, για την περίοδο μετά το 2020. Όπως υπόθηκε ήδη, το καλοκαίρι του χρόνου θα κάνει η Κομισιόν τις προτάσεις της. Έτσι έχουμε 7-8 μήνες μέχρι να κυκλοφορήσουν οι προτάσεις μας. Πρώτο σημείο, η σπουδαιότητα των διαρθρωτικών αλλαγών. Για ποιο λόγο? Διότι όταν αναφερόμαστε σε περιφέρειες που υπολείπονται της ανάπτυξη που είναι λιγότερο αναπτυγμένε, παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ο τομέα των επιχειρήσεων. Όταν κοιτάει κανείς τι λιγότερο αναπτυγμένε περιφέρειες, έχουν λιγότερε επιχειρήσει, μικρότερε επιχειρήσει, μικρότερε ε, ε, νέε επιχειρήσει ε, και, και λιγότερες μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε ένα μη, μη ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι μικρέ επιχείρησεις δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά σε τέτοια περιβάλλοντα, ενώ οι μεγάλε τα καταφέρνουν. Αυτό λοιπόν το μη ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον δεν αποτελεί απλά εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη. Αποτελεί και εμπόδιο για επενδύσει στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στην τωρινή περίοδο επενδύουμε 70 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Αυτές οι επενδύσεις θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασία, μόνο εφόσον το κόστο ίδρυση και ε, λειτουργία μια επιχείρηση δεν είναι υπερβολικά υψηλό, ή μόνο αν οι επιχειρήσει στι εν λόγω περιοχέ έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ ορισμένε δεν έχουν. Για να το πω ε, με δύο λόγια, αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή για το μέλλον είναι πώς μπορούμε να δώσουμε θετικά κίνητρα ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Δείτε για παράδειγμα το επιχειρηματικό περιβάλλον σε αυτές τις περιοχές ώστε να επενδύουμε όχι μόνο σε ανθρώπους και επιχειρήσεις αλλά και στην υπέρβαση των διοικητικών εμποδίων ε, για να πραγματοποιηθούν οι διοικητικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, προσπαθούμε να βρούμε κίνητρα, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα τη λύση. Δεύτερο σημείο, η σπουδαιότητα τη ε, ποιότητα τη διακυβέρνηση. Για μια φορά, αν κοιτάξει κανεί ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη, είναι η αποτελεσματική διαχείριση τη χρηματοδότηση, ε, τη πολιτική συνοχή. Εκεί εστιαζόμαστε στι δημόσιε διοικήσει σε ορισμένα μέρη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη. Εδώ αναφέρομαι στην ποιότητα της ε, δημόσιας διοίκησης, τον έλεγχο της διαφθοράς, ε, την ε, αποτελεσματικότητα του δικαστικού. Είναι σαφές λοιπόν για όλους μας ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις δημόσιες διοικήσεις και τους θεσμούς σε κάθε χώρα για να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη και για να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις χρηματοδοτήσεις. Στο μέλλον λοιπόν θα θελήσουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τον εξυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεων ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές. Τρίτο σημείο, η Επιτροπός μου ήδη ανέφερε ότι η πολιτική συνοχή στο μέλλον θα πρέπει να εστιαστεί σε τομείς υψηλής προσθέμενης αξίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλιματική δράση, κοινωνική ένταξη κτλ. Αλλά μια καλή πολιτική χρειάζεται και έναν καλό μηχανισμό εφαρμογής και εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι μηχανισμοί εφαρμογής ε, τη πολιτική συνοχή έχουν καταστεί πολύ περίπλοκοι. Είπε η Επιτροπός και το επαναλαμβάνω, πραγματικά έχουμε στο νόμο σε αυτή τη στιγμή μελετάμε ριζική απλούστευση. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά το εννοούμε πραγματικά. Αυτό που θέλω να πω είναι και σας το υπόσχομαι εδώ και τώρα ότι ο κανονισμός που θα έρθει στο μέλλον θα είναι πολύ συντομότερος, πολύ απλούστερος, οι κανόνε θα είναι πολύ απλούστεροι θα υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι, λιγότεροι οικονομικοί έλεγχοι, λιγότερες εκθέσεις με στόχο, με το σκεπτικό να βασιζόμαστε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν στους εθνικούς κανόνες και εθνικές αρχές. Όπως τόνισε και η Επίτροπος, αυτό απαιτεί εμπιστοσύνη από όλες τις πλευρές, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Γνωρίζοντας φυσικά ότι η πραγματικότητα πολλές φορές είναι διαφορετική. Θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να το τραβήξουμε όλο αυτό, αλλά πραγματικά πιστέψτε μου, σας δίνω το λόγο μου. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε θετικά αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος γιατί πιστεύω ότι όλοι στην Κομισιόν πλέον συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημερινό πλαίσιο. Το τελευταίο που ήθελα να πω, ε, τα αποτελέσματα της πολιτικής. Ε, ε, ο αντίκτυπος της πολιτικής, θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή, θέλουμε να εστιαστούμε περισσότερο στο μέλλον σε καινοτόμε μορφές χρηματοδότησης. Να απομακρυνθούμε, να εγκαταλείψουμε σιγά σιγά τι επιχορηγήσει και να κινηθούμε προς τα δάνεια, τι εγγυήσει, τα μετοχικά κεφάλαια. Όπως είπε και η κυρία Μιχαήλοβα, αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε ένα τέτοιο πακέτο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση των ε, χρηματοοικονομικών μέσων χρηματοδοτικών μέσων. Συγγνώμη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τι επιχορηγήσει, διότι είναι σαφέ ότι σε ορισμένου τομεί οι επιχορηγήσει είναι η μόνη πηγή χρηματοδότηση για τον απλούστατο λόγο ότι δεν παράγονται έσοδα σε αυτού του τομεί. Οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα άλλα ε, χρηματοδοτικά μέσα μόνο εφόσον υπάρχουν έσοδα. Για μα ε, το σημαντικότερο είναι ότι η πολιτική πρέπει να είναι πρώτη και μετά να ακολουθεί το μέσο το εργαλείο. Τι σημαίνει αυτό, ότι η πολιτική συνοχή δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αφορά ποσοστά χρηματοδότησης, ε, μόχλευση, ε, ποσοστά απόδοσης. Ακόμη και με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, αυτό που μας νοιάζει είναι αν αυξάνουμε την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Αυτό, αυτό θα είναι το μέτρο ε, το οποίο θα λαμβάνουμε υπόψη και όχι τα επίπεδα επένδυση όπως λαμβάνουν υπόψη άλλα εργαλεία διότι λειτουργούμε σε περιοχές, σε αγορές όπου κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Η πολιτική λοιπόν πρέπει να έχει προτεραιότητα σε όλες τις περιπτώσεις. Ήδη τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν μέσω χρηματοδοτικών μέσων και θα βελτιώσουμε, πιστεύουμε, τη χρήση του στο μέλλον. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν μιλήσατε για την απλούστευση, άκουσα την αντίδραση και ε, των συμμετοχόντων είναι η γνωστή αγαπημένη διαδικασία. Ξέρουμε ότι κάθε απλούστευση περνάει πρώτα από πιο περίπλοκες διαδικασίες. Ελπίζουμε όμως ότι αυτή τη φορά οι προσπάθειές μας θα ε, βρουν μεγαλύτερη επιτυχία. Με μεγάλη μου χαρά θα δώσω το λόγο στον ε, επόμενο μιλητή, την επόμενη Επιτρέψτε να το κάνω στα βουλγαρικά. Ευχαριστούμε, λέει η κυρία Βασίλεβα. εξωτήμα μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Επιτροπή Περιφερειών, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτό το σημαντικό φόρουμ ω εκπρόσωπο του Βουλγαρικού ε, Κοινοβουλίου για να σα ε, παρουσιάσω την εμπειρία και το όραμα τη Βουλγαρίας για το μέλλον τη πολιτική συνοχή μετά το 2020. Και τώρα θα περάσω στη μητρική μου. Φέτος κλείνουμε τα 10 χρόνια από την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε λίγο θα αναλάβουμε και για πρώτη φορά την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δέκα χρόνια μετά την ένταξή μας ε, στη Βουλγαρία παραμένουμε ε, τρομερά αισιόδοξοι σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια δημοσκόπηση που έγινε στη Βουλγαρία ε, φάνηκε ότι το 50% των πολιτών στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 63% τη βλέπουν ως δημοκρατική και 52% τη θεωρούν μια ένωση αλληλεγγύης και προστασίας. Σε μεγάλο βαθμό, αυτές ε, οι απόψεις οφείλονται στην πολιτική συνοχή που είναι ε, βασική σημασία για την Ευρώπη. Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής αυτής θα συνεχιστεί και θα αποτελέσει τμήμα των προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας, Αναμένουμε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το 2018 που θα, ε, θα είναι η απαρχή μιας ε, ευρύτερης συζήτησης και γύρω διαβουλεύσεων. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε και πίσω προς το παρελθόν. Μιλώ για την πολιτική συνοχή σε μεγάλο βαθμό βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τώρα ως ε, μέλος του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου. Έχουμε πολύτιμη εμπειρία σε σχέση με το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το περιβάλλον για την περίοδο 2007-2013. Από ένα πρόγραμμα το οποίο βρισκόταν σε κίνδυνο και αναστολή χρηματοδότησης για σχεδόν ένα χρόνο, ε, περάσαμε σε ένα success story παρά τις ε, δυσκολίες δημιουργήθηκε μία σειρά νέων σύγχρονων δομών. Εξυγχρονίσαμε 2.600 χιλιόμετρα ε, ε, και αρδευτικών συστημάτων. Όλα αυτά έχουν ε, ε, ωφελήσει πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες. Τα αποτελέσματα για την Βουλγαρία για την περίοδο 2007-2013 είναι εξαιρετικά θετικά. Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης ήταν 98%, σχεδόν 15 δις λιγότερα. Αυτά είναι μόνο τα στοιχεία, όμως ε, ο αντίκτυπος είναι προφανής και ορατός προς όλους τους Βουλγαρούς πολίτες. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι εξαιρετικά σημαντικά για την βουλγαρική οικονομία και τα ωφέλη ε, γίνονται προφανή αν συγκρίνουμε και τα μακροοικονομικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και το προθετικό σενάριο που δεν θα υπήρχε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Βάσει μιας οικονομετρικής μελέτης της δεκαετούς μας ε, συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΑΕΠ της χώρας μας είναι 10% πάνω και οι εξαγωγές ε, πάλι πάνω από 6% παραπάνω σε σχέση με την έλλειψη ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Έχουν δημιουργηθεί 372.000 θέσεις απασχόλησης. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 9,6% σε σχέση με ένα σενάριο χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ευρωπαϊκέ επενδύσει περιορίζουν τον αρνητικό αντίκτυπο τη οικονομική κρίση. Η Βουλγαρία είναι οικονομικά σταθερή χώρα. με χαμηλά επίπεδα ανεργίας 6,5% και 1% αύξηση στα εισοδήματα, ιδίω ε, σε συγκεκριμένου τομεί. Η πραγματική περίοδος 2014-2020 έδωσε μεγάλη έμφαση στο στρατηγικό χαρακτήρα των επενδύσεων. Η εισαγωγή της ε, αιρεσιμότητας ε, συνδέθηκε με πολλές μεταρρυθμίσεις. Πράγματι, στην αρχή είχαμε κάποιες καθυστερήσεις εξαιτίας των καθυστερήσεων των νομοθετικών δεσμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάστηκε και ένα διάστημα προσαρμογή στους νέους κανόνες. Ε, παρ' όλα αυτά είμαστε 7 στα επίπεδα πληρωμών για τον Οκτώβριο βάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς ε, βλέπουμε τα επόμενα βήματα μετά το 2020. Μπροστά μας έχουμε πολλές προκλήσεις, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Brexit, ε, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πετύχουμε οικονομική ευημερία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει βασικός παγκόσμιος ε, φορέας. Τα βασικά μας μενήματα είναι σύγκληση, απλούστευση, ευελιξία και αυτά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να συνεχίσουμε τον μακρόπνο σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής. Παρά τις αλλαγές πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και να παραμείνει προτεραιότητα στο γενικό προπολογισμό της Ένωσης και μετά το 2020. Χάρη σε αυτή την πολιτική ε, προάγεται η σύγκληση και τα αντιμετωπίζονται διαφορετικά προβλήματα σε όλες τις περιφέρειες. Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ο χρόνος. Γι' αυτό και θα πρέπει να προετοιμάσουμε το νομοθετικό πλαίσιο εγκαίρως και ε, να εφαρμόζονται οι αλλαγές σταδιακά για να μην έχουμε καθυστερήσεις. Το σημαντικό για τη Βουλγαρία είναι να επικεντρωθούμε σε αυτή τη συζήτηση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ακτικού των επενδύσεων προ όφελο τη ενιαία αγορά. Αυτό είναι επωφελέ για όλου. Και έτσι αναπτύσσεται και, οι και μικρές οικονομίες, αλλά και οι χώρες που είναι καθαροί χορηγοί. γιατί βλέπουμε ότι τελικά οι επενδύσεις αυτές προς τις μικρές οικονομίες επιστρέφουν ως κέρδος και ως όφελος στις οικονομίες των δυτικών ε, ευρωπαϊκών χωρών. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από τον έλεγχο και την συμμόρφωση και, τον... Ε, και τα έγγραφα θα πρέπει να περάσουμε σε ένα... μια ιδιαίτερη έμφαση προς τα αποτελέσματα. Βέβαια, ε, πάντα με σεβασμό προς ε, τους κανόνες της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης. Υπάρχουν πολύ υψηλά επίπεδα ελέγχου και λογοδοσίας. Γι' αυτό θα πρέπει να εισαχθεί η αρχή του άπαξ ελέγχου, Single Audit Principle. Εμάς μας ε, ε, απασχολεί αυτό κυρίως σε ό,τι αφορά και τα ταμεία από την πολιτική συνοχής. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στα, στη θέσπιση προγραμμάτων, την εκτέλεση και τον έλεγχο. Πρέπει να συζητήσουμε επίσης το θέμα της ε, αύξησης της οριοθέτησης μεταξύ των ε, ταμείων και κονδυλίων και να αναπτύξουμε ολοκληρωμένες επενδύσεις βάσει στρατηγικής. Χρειαζόμαστε ψηλά επίπεδα ευελιξής για να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένε προκλήσει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υλοποιήσουμε ευέλικτου ε, συνδυασμού ε, προγραμμάτων και εργαλείων, για παράδειγμα ορίζουν 2020 και πρόγραμμα για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με την εναρμόνιση των κανόνων για τα κεντρικά προγράμματα και τα ευρωπαϊκά διευθυντικά και επενδυτικά ταμεία. Κατά την πρώτη προγραμματική περίοδο εμείς οικοδομήσαμε ικανότητες ε, σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Jessica, το Jasper και το Jeremy ήταν ε, θετικά παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση. Όμως και τα καλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ε, τις επιδοτήσεις. Θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά σε συγκεκριμένους κανόνες, μάλλον τομείς τη αγοράς. Τέλος, ενισχύεται η ευθύνη των κρατών μελών και συμβάλλουμε έτσι στην ε, ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων φορέων. Γιατί έτσι ε, τους μαθαίνουμε καλύτερη εκπαίδευση με καλύτερο σχεδιασμό και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την αρχή της θεματικής συγκέντρωσης για την επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Ελπίζω η αιρεσιμότητα να ενισχυθεί περαιτέρω και μετά το 2020. Για τις κυρώσεις όμως, πέρα από τις κυρώσεις πρέπει να έχουμε όμως και κίνητρα. Στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο ε, έχουμε και ένα μότο μπροστά που λέει ισχύσει εν τη ενώση». Αυτό θα είναι και το μότο της Βουλγαρικής Προεδρίας. Πιστεύω ότι με τις κοινέ προσπάθειες έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και ελπίζω με τη συζήτηση που θα γίνει ε, να καταφέρουμε να αυξήσουμε τη συνεργασία μας για περισσότερη Ευρώπη και για μια ευφυή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής. Ε, Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δίνω το λόγο στην κυρία Ροβάνα Πλάμ, πρόεδρο τη Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, του Κοινοβουλίου τη Ρουμανία. Έχετε το λόγο, κυρία Πλάμ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Μιχαήλοβα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που μας προσφέρετε σήμερα να έρθουμε εδώ και να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020. Αφορά το δικό μας μέλλον το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το μέλλον όλων μας, όλων των Ευρωπαίων. Σήμερα θα σας μιλήσω και υπό τις δυο μου ιδιότητες ως ε, πρώην ε, υπουργό Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και ε, ως σήμερα, όπως είπατε, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Κοινοβουλίο της Ρουμανίας, αλλά και ως εκπρόσωπος της Ρουμανίας η οποία θα αναλάβει την Προεδρία το πρώτο του 2019. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο από το 2007 μέχρι το 2013. Αυτή η περίοδος για τη Ρουμανία από το 2007 μέχρι το 2013 υπήρξε η πρώτη εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε εκείνη την περίοδο μαθαίναμε, κάναμε λάθη, αλλά καταφέραμε και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της χώρας. Οι παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής ε, μας έδειξαν την προσθέμενη αξία της πολιτικής. Αν πάρουμε ως παράδειγμα το αποτέλεσμα μόχλευσης ε, των κονδυλίων, κάθε ευρώ που δαπανήθηκε οδήγησε σε αύξηση του ΑΕΠ συσσωρευμένη των 2,3 ευρώ στη Ρουμανία. Το ποσοστό απορρόφησης ήταν περίπου 90% στο τέλος περίοδου. Η περίοδος 2014-2017 ε, Εκεί απλουστεύσαμε περισσότερο και εστιαστήκαμε περισσότερο στα αποτελέσματα. Εκεί ε, εισήχθηκε η εξάντερεσιμότητα. Ωστόσο, οι κανόνε εκείνη περίοδου ήταν πιο περίπλοκοι υπήρχαν και περισσότερε κατευθυντήρε γραμμέ από ό,τι στην προηγούμενη περίοδο. Αυτό σε συνδυασμό με την καθυστέρηση τη υιοθέτηση των κανονισμών πολιτική συνοχή καθυστέρησαν την έναρξη τη εφαρμογή. Ήθελα επίση να επισημάνω ότι ο προγραμματισμό είναι δυσκολότερο όταν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένα κατόφλια που ορίζονται σε κεντρικό επίπεδο χωρί να λαμβάνονται υπόψη επενδυτικέ ανάγκε όλων των κρατών μελών και περιφερειών. Το μέλλον της πολιτικής συνοχής σχετίζεται στενά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπα. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Εξακολουθούμε, να χρειαζόμαστε μια ισχυρή, δυνατή ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής ε, για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ώστε να γεννηθεί έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία. Αυτή η πολιτική πρέπει να διατηρεί το ρόλο τη ω η σημαντικότερη ευρωπαϊκή επενδυτική πολιτική. Θα πρέπει να δημιουργεί ολοκληρωμένε λύσει προσαρμοσμένε ε, στι ευρωπαϊκέ, εθνικέ, περιφερειακέ και τοπικέ απαιτήσει, λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε των, ανθρώπων ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου να επισημάνω ορισμένα προβλήματα για το μέλλον τη πολιτική συνοχή ε, μετά το 2020, που θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιληθούν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πρώτα απ' όλα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της χρήση των κονδυλίων. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέε προκλήσει και προτεραιότητε όπω η ασφάλεια, οι μετανάστε και τα σύνορα, πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να εστιαστεί στι πραγματικέ ανάγκε που έχουν ε, εντοπιστεί σε επίπεδο περιφερειών και θα πρέπει να διατηρηθεί και το επίπεδο των ε, πιστώσεων σε, για αυτές τις ανάγκες. Θα πρέπει να εντείνουμε την αποτελεσματικότητα λοιπόν χρήση των κονδυλίων. Δεύτερον, έξυπνη μετάβαση μεταξύ προγραμματικών περίοδων. Κάθε νέα περίοδος ε, έφερε νέες ιδέες αλλά δημιούργησε και επιπλοκές. Πάντα πρέπει να καθορίζουμε το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου με νέες διαδικασίες και κανόνες. Οι κατευθυντές γραμμές ε, της Κομισιόν καθυστερούν και συμπληρώνουν απλά τους εθνικούς κανόνες. Συνεπώς, η Κομισιόν θα πρέπει να σκεφτεί στο μέλλον πώς να διατηρήσει τις τρέχουσες δομές. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις υπάρχουσες δομές και όχι να ξαναξεκινάμε ε, διαπίστευση κάθε νέα περίοδο ε, για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τρία, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις πραγματικές ανάγκες των περιφερειών και των κρατών μελών. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τη χρηματοδότηση του σημερινού κανονισμού ERDF για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία, ICT και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την κυκλική οικονομία. Οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη θα πρέπει, πιστεύω, να αναπτύξουν επενδυτικές στρατηγικές ε, και να βασιστούν στο ότι μπορούν να εντοπίσουν ποιε είναι οι προτεραιότητε που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τα διάφορα διαθέσιμα κονδύλια. Αυτό θα βοηθήσει τα κρατημέλη και τις περιφέρειες να αρχίσουν να εντοπίζουν τις ανάγκες και στη συνέχεια να αναζητούν τη σωστή πηγή χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι οποιοδήποτε κατόφλιο το οποίο ε, εκπονείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το μερίδιο ESF δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη σωστή ε, κατανομή μεταξύ προτεραιοτήτων ESF και ERDF που θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό ε, και κρατικό επίπεδο. Τέσσερα, συνδυασμός ε, χρηματοδοτικών μέσων με επιχορηγήσεις. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι σημαντικά τα χρηματοδοτικά μέσα και ότι μπορούν να ε, βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη μαζί με τις επιχορηγήσεις. Η Ρουμανία θεωρεί ότι έχουν ύψιστη σημασία στην περίπτωση έργων που δημιουργούν εισοδήματα. Συμπληρώνουν τα κονδύλια, τα διαρθρωτικά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε το σύστημα χρηματοδότηση που βασίζεται σε επιχορηγήσει. 5. Η σύνδεση μεταξύ πολιτική συνοχή και ευρωπαϊκού εξαμήνου. Οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει είναι σημαντικέ και θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για μια ορθή πολιτική συνοχή. Η σύνδεση μεταξύ πολιτική συνοχή και ευρωπαϊκού εξαμήνου θα πρέπει να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί. Ωστόσο, οι συστάσει αναχώρα θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμες και να συμπεριλαμβάνουν μηχανισμούς κινήτρων αντί για κυρώσεις ή αιρεσιμότητα. Κατά την άποψή μας, οποιοδήποτε διορθωτικό μέτρο δεν θα είναι παραγωγικό, δεν θα βοηθήσει να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στις συστάσεις αναχώρα. Θα πρέπει να εστιαστούμε σε αυτές τις συστάσεις αναχώρα, που είναι σημαντικέ στον τομέα τη πολιτική συνοχή και να θα πρέπει να βοηθήσουμε να παγιωθεί το επενδυτικό πλαίσιο. Έξι, απλούστευση και ευελιξία για τους δικαιούχου. Η Ρουμανία υποστηρίζει την πρόταση δημιουργία ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για όλα τα κονδύλια και την ευθυγράμμιση των κανόνων για όλα τα ταμεία με προγράμματα ή έργα ίδιου τύπου. Όλα αυτά πιστεύουμε θα συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πόρων. Μαζί με αυτό υποστηρίζουμε την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίηση, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές και οι δικαιούχοι. Κατά την άποψή μας είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των στόχων της απλούστευσης ασφάλειας και επιδόσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν οι κανονισμοί όσον αφορά για παράδειγμα την συγκέντρωση των θεμάτων, τους κανόνες ε, οικονομικών και λοιπόν ελέγχων, της αιρεσιμότητας εξάντε, ε, της καθιέρωσης δικτών, ε, επιλογών, απλοποιημένων επιλογών κόστους κτλ. Επιπλέον, όσον αφορά την ευελιξία, πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη, ώστε να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στις νέες προκλήσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τη στρατηγική κατεύθυνση και τη βεβαιότητα των προγραμματικών εγγράφων, τα οποία είναι πολιτή. Οποιαδήποτε λύση εδώ μπορεί να βοηθήσει σε απρόβλεπτες δράσεις ε, ε, με εξαίρεση από τον ε, κανόνα θεματικής συγκέντρωσης και που θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΣΥΦ. Επίση, κατά την άποψή μας, πρέπει να είμαστε και πιο ευέλικτοι στον καθορισμό των τομέων που θα χρηματοδοτούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητα, ώστε να προσδιορίζεται μια πραγματική σύγκληση και ε, ε, ισορροπημένη ανάπτυξη των κρατών και των περιφερειών και τη Ευρώπη στο συνολό το να αυξηθεί η αμοιβή εμπιστοσύνη των βασικών παραγόντων που εμπλέκονται στην υλοποίηση τη πολιτική συνοχή. Αυτό ο στόχο θα πρέπει να είναι μια από τι αρχέ τη πολιτική συνοχή, με στόχο να ενισχυθεί η αμοιβή εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των βασικών παραγόντων, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τη πολιτική μέχρι την υλοποίηση, ώστε να αποφεύγεται ε, υπερβο... κανονιστικό υπερθεματισμό και πολλαπλασιασμό των ε, ε, ελέγχων και υπερβολική υπερβολικές ρυθμίσεις. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο υλοποίησης, οι απόψεις εδώ δίστανται. Άλλοι υποστηρίζουν 7 ετία, άλλοι 5 ή πέντε συν 5. Εγώ πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να πλουστεύσουμε τους κανόνες και να ξεκινήσουμε τη χρηματοδότηση δικαιούχων από την ημέρα 1 της περίοδου, μπορούμε να προβλέψουμε το διάρκεια του επόμενου ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020. Ωστόσο, η Ρουμανία είναι υπέρ του να διατηρηθεί επταετή περίοδο λόγω τη ε, σπουδαιότητα ε, τη διατήρηση του στρατηγικού χαρακτήρα του προπολογισμού ω σταθερού και προβλέψιμου εργαλείου για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, θα ήθελα να πω ότι η Ρουμανία θα συντονιστεί με τι Προεδρίε Βουλγαρία και Αυστρία και θα εργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υποστηρίξει την έγκυρη υιοθέτηση της πολιτικής συνοχής και των σχετικών κανονισμών πριν από τις εκλογές του 2019. Κάτι που θεωρώ θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα να επισημάνω ότι θα πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε η πολιτική συνοχή να αποτελέσει το κύριο εργαλείο παγίωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ειδικότερα υπό τις σημερινές συνθήκες ευρωσκεπτικισμού. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Πλάμ. Εγώ τώρα έχω κύριο Σνάιντερ που είναι μέλης Επιτροπής των Περιφερειών για να ακούσουμε τώρα και τι λένε οι περιφέρειες οι ευρωπαϊκές για το μέλος πολιτικής συνοχής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ξέρω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών εκτιμά ιδιαίτερα αυτή την πρόσκληση και είναι πάρα πολύ θετικό που συναντώμεθα εδώ και με προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ελπίζω την επόμενη διετία να ε, ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία αυτή. Είπατε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών το Μάιο ε, εξέδωσε μια γνωμοδότηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ε, 350 ψήφοι ε, και η μία μόνο ήταν η ψήφος κατά, άρα βλέπετε ποια είναι η άποψη ε, των αρχών της ε, περιφερειακής τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα σας ε, δώσω κάποιες βασικές ε, σκέψεις, ε, κάποια βασικά σημεία της γνωμοδότησης. Δεν θα ήθελα να επικαλύψω τις προηγούμενες παρεμβάσεις, γιατί τα περισσότερα από όσα υπόθηκαν βρίσκονται στην γνωμοδότηση και με κάνει ιδιαίτερη ευτυχία αυτό, γιατί δεν θα ήθελα να υπάρχουν επίμαχα σημεία, αλλά δεν θέλω να τα επαναλάβω και όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική συνοχή δεν είναι είδο δώρου ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη, στις ε, κοινότητες και στους δήμους, αλλά είναι μια υποχρέωση που πορεύει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, είναι ένα μάστι, είναι μια υποχρέωση αυτή η εδαφική ε, και η κοινωνική συνοχή που πρέπει να ενισχυθεί. Γι' αυτό χρειάζεται και η πολιτική συνοχή. Επομένως, είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει σχετική υποχρέωση που προβλέπεται στις συνθήκες. Όποιος θέλει τώρα να βρει απαντήσει ε, Τι απαντήσεις θα τι βρει στην 7η έκθεση συνοχή, ε, που πολύ καλά λέει ε, πώ θα πρέπει να σκεφτούμε την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Βέβαια αυτή η πολιτική συνοχή όπω είναι σήμερα δεν είναι τέλεια βέβαια. Υπάρχουν τεράστιε ανάγκε βελτίωση και αυτό έχει να κάνει και με μονομένε τεχνικέ πτυχέ που δεν θέλω τώρα να αναφέρω αναλυτικά αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί για να είναι πιο αποτελεσματική. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματική αποτελεσματικότητα τη Και όπω είπε και ένα από τους προλαλήσαντες ομιλητέ, πρέπει να υπάρξει απλούστευση. Ο κύριο ε, Φονμπρέσκα ήταν αυτό που το είπε πραγματικά πάρα πολύ ξεκάθαρα. Πρέπει να υπάρξει απλούστευση. Όταν άρχισα εγώ να προετοιμάζω αυτήν την ε, νομοδότης από την Επιτροπή ε, Συνοχής, στις πρώτες σκέψεις μου ήταν ότι το θέμα που θα χαρακτηρίσει τα επόμενα χρόνια είναι η λέξη απλούστευση ε, και χαίρομαι που υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από όλες τις πλευρές αλλά δεν χαίρομαι γιατί φαίνεται ότι είναι και παντού υπαρκτό αυτό το πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει σίγουρα μεσοπρόθεσμα ε, να ε, βελτιώσουμε αυτή την αποτελεσματικότητα και αν δεν υπάρξει απλούστευση οι προσπάθειές μας θα πέσουν στο κενό. Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική συνοχή. Αν δεν έχει τα απαραίτητα μέσα, το απαραίτητο προπολογισμό δεν πρόκειται να επιτύχει και θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη ε, στις, ε, στον προβληματισμό μα. Ε, δηλαδή να δούμε την πρικοδότηση, όχι σε απόλυτα νούμερα, αλλά αναλογικά πώ είναι σήμερα και έτσι πρέπει να συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε βελτίωση, αλλά όχι και καμία άρδιν ανανέωση της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, ε, εκεί που εφαρμόζονται δηλαδή τα σχετικά, υπάρχει προειδοποίηση. Ναι, προσέξτε, σίγουρα να υπάρξει ανακαίνιση, θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση και απλούστευση, αλλά μην αλλάξετε πάρα πολλά, γιατί ε, αυτοί που πρέπει να εφαρμόσουν επιτόπου, ε, οι αρχές τοπικής αυτοδικής θα βρεθούν όπως το 2014 σε, μπροστά σε ένα τεράστιο όγκο νομοθετημάτων και δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν ε, ε, είναι πάρα πολύ υπερβολικό το βάρος ε, και για τους, τις και για τους δικαιούχους. Στο μέλλον η πολιτική συνοχή πρέπει να παραμείνει προσφόρα προς όλες τους Δήμους και Περιφέρειες και θέλω να σας ευχαριστήσω που το είπατε, οι προλαλήσαντες θα την αποδεχθούν όλοι την πολιτική συνοχή μόνο αν επί της αρχής αφορά και προορίζεται για όλες τις περιφέρειες. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, αλλά βασικά αυτό πρέπει να παραμείνει η προσφορά να μην αλλάξει. Η αρχιτεκτονική τώρα, δηλαδή η κατανομή σε διάφορες ε, ε, κατηγορίες, δεν νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξει, έχει αποδείξει την αξία της ε, η μέχρι τώρα κατηγοριοποίηση ε, και σίγουρα υπάρχουν ε, κάποια αναπτυξιακές κατηγορίες και αν δει κανείς ε, τη συμμετοχή και την κατανομή βλέπει τις ομοιότητες μεταξύ των περιφέρουν που ανήκουν στις ε, κατηγορίες και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουν αυτές οι κατηγορίες. Φυσικά ένα άλλο θέμα που συστήθηκε είναι ε, τα κριτήρια ε, του ΑΕΠ, αν θα πρέπει το κριτήριο του ΑΕΠ να παραμείνει. Και θεωρούν τα κρατη ότι πρέπει να παραμείνουν ένα αποφασιστικό κριτήριο για την κατηγοριοποίηση των περιφερειών. Ωστόσο, υπάρχει άποψη ότι πρόσθετα κριτήρια θα πρέπει να προταθούν. Δηλαδή να πάμε σε ένα πιο βαθύ επίπεδο για να δούμε συγκεκριμένα εντό των κρατών μελών πώ κατανέμονται τα κονδύλια συνοχή. Σίγουρα υπάρχουν δείκτε που έχουν το ρόλο και σήμερα θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά και νομίζω να προσθέσουμε νέου δείκτε. Ένα σημαντικό ακόμη θέμα είναι ε, ποια είναι η σχέση μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων σε ό,τι αφορά ε, την διαχείριση ε, των ε, κονδυλίων με την κεντρική διαχείριση. Εμείς θεωρούμε και απευθύνουμε σχετικά έκκληση αυτό που πρέπει να γίνει να μην υπάρχει μια αντίθεση και μια αντιπαράθεση και τα δύο είναι δικαιολογημένα. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί είναι η συνέργεια, είναι η αλληλεπίδραση των μεθόδων και της χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σίγουρα εδώ περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν υπάρχουν. Πιστεύουμε ότι σε ό,τι αφορά ε, την χρησιμοποίηση των ε, διατεθέντων κονδυλίων, δηλαδή των κονδυλίων συνοχής, πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Ε, τα είπε ξεκάθαρα και επίτροπε, επίτροπος. Πρέπει να υπάρξει ευελιξία. Αυτό σημαίνει ενίσχυση επιτόπου της εδαφικής διαχείρισης. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο τοπικό επίπεδο, γιατί οι τοπικές αρχές ξέρουν τι είναι καλύτερο. Δεν μπορούν να αποφάσουν να λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο το λέω αυτό βέβαια και ταυτόχρονα απευθύνω έκκληση και στα κράτη-μέλη, γιατί δεν μιλάω μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά Απευθύνω έκκληση και στα κράτη-μέλη να εμπιστευτούν περισσότερο τις, περιφέρειες και να μην αφαιρούν αρμοδιότητες από τις περιφέρειες. Αυτό το θέλω να το πω ξεκάθαρα. Επίσης το θέμα των ερεσιμοτήτων, ε, τα conditionalities, όρων και προϋποθέσεων, τα συμφωνήσαμε και συμφωνούμε στην Επιτροπή ε, των Περιφερειών ότι ε, δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο. Ερεσιμότητα δεν ταιριάζει με πολιτική συνοχή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται, που θα είναι κοινωνικά, οικονομικά, κοινωνική, οικονομική, εδαφική συνοχή. Αυτά είναι τα σχετικά κριτήρια και ανάλογα με τις ανάγκες. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια εκτός πολιτικής συνοχής, αλλά μόνο εντός πολιτικής συνοχής. Ε, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται η Επιτροπή αυτή να επιτύχει. Το λέμε και είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Επομένως, αιρεσιμότητες, ε, εκφράζουμε την επιφυλακτικότητά μας. Επίσης, σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και διαθροτικών ταμείων. Πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η σχέση. Φυσικά, βλέπουμε στην πρακτική κάπως ε, να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά περιθώρια ε, βελτιώσεων υπάρχουν ακόμη πολλά. Και οι περιφέρειες ε, θα πρέπει να συμμετάσχουν ε, πιο ενεργά και πιο στενά στις συζητήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, γιατί πολλές φορές δεν αναφέρονται στα αιτήσια πράγματα, προγράμματα ή συστάσεις αναχώρα. Είναι σχεδόν διαφορετικοί κόσμοι, αλλά εμείς πρέπει αυτά να τα φέρουμε πιο κοντά. Και επειδή τελειώνει σιγά σιγά, σιγά ο χρόνος έχω δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η σημερινή συνάντηση και σας παρακαλώ να μην είναι μία και μόνη αυτή η συνάντηση απάντηση ε, το 2020 ξεκινάει η νέα περίοδος προγραμματισμού. Το Μάιο του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα θα καταθέσει την πρότασή της Κομισιόν για το προσεχές πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κράτη-μέλη ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια θα λάβουν την απόφαση. Τα κοινοβούλια θα αποφασίσουν. Εμείς εδώ λοιπόν όλοι που είμαστε φίλοι της συνοχής, της πολιτικής συνοχής, τέλος πάντων μας αφορά η πολιτική συνοχή, το λιγότερο που μπορώ να πω, είναι πολύ καλό να ε, συνεδριάζουμε από κοινού. Τώρα, στην Επιτροπή των Περιφερειών τον Μάιο ε, δημιουργήσαμε ένα, μία ένωση που τη λέμε Cohesion Alliance, Συμμαχία για τη Συνοχή. Και Όλοι μπορούν να είναι μέλη, είτε μεμονωμένοι ιδιώτες, είτε μέλη ε, κυβερνήσεων, κοινοβουλίων εθνικών, ευρωπαϊκού, οποιοδήποτε. Κυρίες και κύριοι, ορίστε, το hashtag στο Twitter ε, μπορείτε ήδη να πάτε και να γίνετε μέλος. Cohesion Alliance, μία λέξη, βλέπετε. Έχουμε χιλιάδες και όσο περισσότερες χιλιάδες έχουμε τόσο πιο ισχυρή θα γίνει αυτή η συμμαχία, αυτός ο συνασπισμός και τόσο περισσότερο θα επηρεάσει τις μελλοντικές συζήτησεις. Ευχαριστώ και παρακαλώ γίνετε μέλη. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Ελπίζω να έχουμε όλο και περισσότερους ε, υποστηρικτές ε, τέτοιων πρωτοβουλειών, όπως η Συμμαχία για τη Συνοχή. Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των Open Days για τις πόλεις και περιφέρειες και ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών. Σας ευχαριστούμε. Προχωρούμε τώρα με την κυρία Κρέο. Είναι μέλος της Επιτροπής Ρέτζη και εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τι να πει κανεί σε δέκα λεπτά, δεν μπορεί βέβαια σε καμία περίπτωση να πραγματευτεί την πολιτική συνοχή, ούτε καν το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Γι' αυτό θα περιοριστώ και εγώ σε λίγα και μόνο σημεία. Πρώτα απ' όλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μα Επιτροπή εδώ και πολλού μήνε ε, συζητά ε, το μέλλον τη πολιτική συνοχή. και πραγματικά, ε, η, όπως το γνωρίζετε και εσείς, φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προωθήσει μια ε, πολιτική συνοχή στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες και αυτές που έχουν την λιγότερη ανάπτυξη και αυτές που έχουν την περισσότερη ανάπτυξη και αυτές που είναι κάπου σε μεταβατική φάση. Διότι είμαστε βέβαιοι ότι το εργαλείο αυτό της πολιτικής συνοχής δεν είναι μόνο ε, ένα μέσο επενδύσεων για το σύνολο της Ένωσης, αλλά είναι και μια έκφραση αλληλεγγύης για τις περιφέρειες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια προϋπόθεση για όλα αυτά και θα ήθελα να το πω ίσως λίγο πιο ξεκάθαρα από τον προλαλήσαντα φίλο προϋπόθεση είναι να υπάρχουν επαρκή σπόροι, επαρκή χρηματοδότηση. Και το λέω απερίφραστη και ξεκάθαρη. η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί από τη μία πλευρά όταν ε, χάσει το δεύτερο πιο μεγάλο καθαρό εισφορέα να μείνει με τρύπε στον προπολογισμό και μετά άλλα θέματα που είναι πολύ σημαντικά όπως είναι το μεταναστευτικό ρεύμα, ε, η κλιματική αλλαγή, η νέα πολιτική για την άμυνα, την ασφάλεια και πάρα πολλά πολλά άλλα ε, να τα αναλαμβάνει ως ευθύνε χωρίς τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό προπλασμό ή να δεχθούν ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Εμείς μία φορά μπορούμε να δαπανίσουμε τα ευρώ που έχουμε, όχι πέντε φορές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι ακριβώς με την πολιτική συνοχή ε, για τα ευρώ, το ένα ευρώ, ε, να οργανώσουμε άλλα τέσσερα ευρώ αν θέλετε. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και επειδή εδώ είναι και βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε ότι από κοινού πρέπει να αγωνιστούμε και στα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε τα κράτη-μέλη να δείξουν αυτή την ετοιμότητα και όχι να τα λένε μόνο ε, μεγαλόστομα σε ειδικέ ε, εκδηλώσεις, πανηγυρικές συνεδριάς κτλ. Αλλά θα πρέπει τους υπουργούς οικονομικών τους και όχι μόνο ε, την Ευρώπη να πείσουν ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε το θέμα αυτό παρουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων. αρχή πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερος υπέρ του να έχουμε λίγες αλλαγές ε, στην ε, διάταξη, αν θέλετε, της πολιτικής Όχι να ξεκινήσουμε από την αρχή και να ξαναχρειαστεί να τα μάθουμε από την αρχή τα πράγματα και να πρέπει και η διοίκηση να τα μάθει ξανά από την αρχή και οι δικαιούχοι το ίδιο γιατί και αυτοί βέβαια είναι άμεσα θυγόμενοι. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο πολύ να διατηρήσουμε το σύστημα ως έχει. Σίγουρα χρειάζεται απλούστευση. Το είπε και η Πρόεδρος ε, ότι έχουμε τη διαδικασία του Omnibus. Ε, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για μια πρώτη απλούστευση και ελπίζω, ελπίζω σήμερα ε, που είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο να καταλήξουμε πράγματι σε συμβιβασμό. Βέβαια, το πράσινο φως το τελευταίο θα πρέπει να δοθεί από τα κράτη-μέλη. Αλλά, αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν θετικά μηνύματα και φαίνεται ότι μάλλον θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ε, συμβιβασμό. Γιατί πραγματικά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό στο δρόμο της απλούστευσης για το Simplified Cost Option, ε, για το Single Audit ε, Αυτά είναι σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως κάτι επίσης ενδιαφέρον και πάντα στο απλές της δικασίας Omnibus είναι ένα πακέτο ορατότητας, ε, προβολής, διαφάνειας, visibility package, ε, είπε η Επίτροπος Κρέτσου στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ δεν ήξερε κανένας ε, ότι έχει δοθεί επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς αυτή είναι μία από τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουμε πολύ καλά πράγματα και δεν τα λέμε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πόσα εκατομμύρια πηγαίνουν στι περιφέρειες ή υπάρχει συγχρηματοδότηση. Ε, ποιοι το ξέρουν ε, στα κράτη-μέλη. Μας λένε μόνο γραφειοκράτες. Μας λένε ότι το μόνο που προκαλούμε είναι κόστος, δαπάνες. Δεν βλέπουν όμως πόσα χρήματα, πόσα κονδύλια διαθέτουμε στις Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη προβολή. Αυτό και μέσω της διαδικασίας του Omnibus ελπίζω να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Και έχουμε καταλήξει σχετικό συμβιβασμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ναι στα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά μόνο όταν αυτό είναι λογικό, εκεί που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχή που πραγματικά ε, χρειάζονται αυτά τα κονδύλια, αυτές τις επιδοτήσεις. Ε, Παραδείγματο χάρη, όταν θέλω να στηρίξω ένα ερευνητικό πρόγραμμα, αυτό παράγει εισόδημα, υπάρχει επιστροφή. Ε, δεν είναι όμως αυτό πάντοτε αληθές. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα ε, σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας, για έρευνα δηλαδή. Θα πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, παραδείγματος χάρη για την αλλαγή του κλίματος και να τους υποστηρίξουμε. Και ε, χρειαζόμαστε επιδόματα, επιχορηγήσεις στο μέλλον για τους τομείς αυτούς. Και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, τα λέει ξεκάθαρα. Τώρα, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Νομίζω ότι ε, σωστά ε, έχουν αναφερθεί. Ε, να δώσω ένα παράδειγμα για την ψηφιοποίηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να της δοθεί στο μέλλον πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από τη μέχρι τώρα. Αλλά θεωρώ τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες ε, θα τα συζητήσουμε πολύ καλά και θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα θέματα. Πρέπει όμως να προσέξουμε το εξή. Πολιτική συνοχή ποτέ δεν ήταν και δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει και στο μέλλον να είναι ε, η πανάκια ή κάτι το οποίο θα αντικαταστήσει τα πάντα, για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Ταμείο Λεγγύης για τις φυσικές καταστροφές. Για περικοπές εργασίας, δραστικές, βασικές απαιτήσεις. Έχουμε το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει και εκεί να υπάρξουν απλουστεύσεις και οι πολίτες να μπορούν ε, να αξιοποιούν τα κονδύλια και αυτών των ταμείων. Θα πρέπει εμείς να εστιάσουμε στις δικές μας υποχρεώσεις, δηλαδή στην οικονομική, κοινωνική και αδαφική συνοχή. Δεν πάνε όλα μέσα ε, σε αυτό το, το καλάθι, αν μπορώ να το πω έτσι. Πρέπει να εστιάσουμε στις δικές μας υποχρεώσεις. Υπάρχουν άλλα ταμεία για άλλα πράγματα. Και κάτι τελευταίο, για τις αρεσιμότητες τα conditionalities. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τωρινό ε, πλαίσιο ε, της πολιτικής συνοχής, την τωρινή περίοδο προγραμματισμού, αγωνίστηκε ε, ώστε στον τομέα της πολιτικής συνοχής να μην υπάρχει μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Τα λέω γερμανικά, άρα καταλαβαίνετε πόσο αγώνα έχουμε δώσει και έχω δώσει. Δεν είναι απλά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα, έτσι όπως είναι, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Πώς να το κάνουμε. Και γι' αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Έχει νόημα να υπάρχει αιρεσιμότητα στον τομέα της πολιτικής συνοχής ή μήπως θα είχε πολύ περισσότερο νόημα και θα ήταν πολύ πιο λογικό να δούμε ποιε είναι οι προποθέσει, όροι ή αιρεσιμότητε τέλο πάντων που χρειαζόμαστε, τι πρέπει να υποβάλουμε σε όρου και προποθέσει γιατί εδώ μιλάμε για μια πολιτική που πρέπει να βοηθά τι περιφέρειες. Αυτή είναι η αρμοδιότητά της και όχι να τιμωρεί άλλου για λάθη, για παραλήψεις, περιφερειακέ τα κτλ. Νομίζω ότι από κοινού θα πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να βρούμε τι ευκαιρίε και τι δυνατότητε, ε, για ε, να διαμορφώσουμε με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τη μελλοντική πολιτική συνοχή και εν κατακλείδη. Για το χρονοδιάγραμμα μια λέξη θα μου επιτρέψετε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο πριν τις επόμενες ευρωεκλογές να προχωρήσει τόσο ώστε να έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο, τους πρώτους τριμερείς διαλόγους για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Όμως, αυτό σημαίνει όχι να έχουμε μετά από 8-9 μήνες ε, μια πρόταση για τον κανονισμό για την πολιτική συνοχή. Γιατί άκουσα ότι η τελική απόφαση θα μπορούσε να είναι στα τέλη του 2020 για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όχι, από χρόνο το χρειαζόμαστε αυτό το πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ήδη προτάσεις και θα πρέπει, πιστεύω, οι προτάσεις για το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο να γίνουν παράλληλα με τις προτάσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και πραγματικά έγκαιρα να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το 2021 ε, και να έχουν τα ε, κράτη ε, πάρει εκ των προτέρων τις οδηγίες τους και να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς να το πω, ούτε τα κράτη-μέλη χαρακτηρίζονται κάπως, μπορούν να ομφαλοσκοπήσουν ή μπορούν να θεωρήσουν το καθένα σαν ξεχωριστό τομέα. Χρειάζεται συνεργασία. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο από κοινού. Και φυσικά και η Ευρωπαϊκή δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τα κρατημέρια και χωρίς και τις περιφέρειες βέβαια, τις περιφέρειες μας. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη φορά και όταν θα περιγράψουμε το νομικό πλαίσιο για τα προγράμματα, για τα διάφορα σχέδια κτλ αν τα καταφέρουμε και ελπίζω με αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, να, αν δεν πετύχουμε αυτό, θα χαθεί η εμπιστοσύνη ε, στη δημοκρατία. Αλλιώς, αν πετύχουμε όμως αυτή τη δημοκρατία και αυτή την εμπιστοσύνη, θα την αποκαταστήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ όλους ε, τους ε, βασικούς ομιλητές σήμερα για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους αλλά και για την πειθαρχία που επέδειξαν. Βλέπετε ότι είμαστε εντός του χρονικού πλαισίου. Απίστευτο πραγματικά. Ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο τμήμα της συζήτησης του ανοιχτού διαλόγου, όπου τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη και οι προσκεκλημένοι μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Έχω ένα κατάλογο 20 ομιλητών, το οποίο μας επιτρέπει να δώσουμε στον καθένα τρία λεπτά. ως χρονοομιλίας και θα επιμείνω πολύ σε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να δώσουμε το λόγο σε όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Α, 21 τώρα. Εντάξει, θα το θυμάμαι. Ξεκινούμε με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Και εσείς θα πάρετε λόγο ως ε, συντονίστρια, κυρία Μισελ. Ξεκινούμε με ένα συντονιστή, δύο μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων και άλλον συντονιστή μετά και συνεχίζουμε. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Για τρία λεπτά. Θέλω να συμβάλλω κάπως σε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια, πολλά έχουν υποθεί. Το θέμα είναι ο εξυγχρονισμός της πολιτικής μας και να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Κάποιε φορέ μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερα χρήματα. Δεν θέλουμε πάντα περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Αν δείτε λοιπόν κράτη-μέλη, πολλά ούτε καν σαν τους πόρους το 2014, 15, 16, 17. Κάποιοι μόλι τώρα ξεκίνησαν. Και κάποιοι διπλασίασαν, τριπλασίασαν τον αριθμό των κανόνων που φτιάξαμε στην Ένωση. Ας μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό. για τα αποτελέσματα λοιπόν, όχι μόνο το τι δίνουμε αλλά και τι παίρνουμε. Μετά για την ευελιξία. Ναι, πράγματι θέλουμε κάτι κομμένο και ραμμένο στα χέρια μας ε, και να κάνουμε πολύ περισσότερα να συμφωνήσουμε από αυτού. Αλλά όπω είπε η κυρία Κρέλ, είναι πολύ επίπεδη διακυβέρνηση. Ο επιμερισμός των αποτελεσμάτων και των δικαιούχων. Αυτό είπε και η Επίτροπο. Δείτε τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά, που δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, καμία προβολή του ευρωπαϊκού έργου. Πού ζούμε, στην Ευρώπη δεν ζούμε. Όταν τα κράτη-μέλη λοιπόν ζητούν ευρωπαϊκή ψωθεμένη αξία, αυτό θα πρέπει να προβάλλεται επίσης. Στο Brexit κανείς δεν είπε ότι δεν ήταν το Λονδίνο που μας επέτρεψε να μετατρέψουμε την πόλη μας σε κάτι καλύτερο, αλλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε και με τη νέα πρόταση όμνιμπους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Το ΕΛΚΑ έκανε αυτή την πρόταση. Ας την αφήσουμε λοιπόν να λάμψει. Γιατί αυτό θέλουμε, να συμμετάσχουν και οι πολίτες. Μια εταιρική σχέση. Υπάρχουν τόσα καλά αποτελέσματα που μπορούμε να προβάλλουμε. Όχι μόνο για την δαπάνηση των κονδυλίων, αλλά και μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος όταν έχουμε νέες startup ή καινοτόμες τεχνολογίες ε, στην υγειονομική περίθαλψη, στην κινητικότητα και αλλού. Όχι μόνο λοιπόν να μιλούμε για τα κονδύλια, αλλά και για τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα κονδύλια στην κοινωνία. Δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι οι θεσμοί και οι άνθρωποι θα μας ακολουθήσουν. Όχι, οι ψηφοφόροι ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Και τώρα έχουμε και την πρόταση όμνιμπους και την ενδιάμεσα αναθεώρηση. Κάτι άλλο τώρα. Α εξετάσουμε την ταχεία διαδικασία. 5% των κοντιλίων να τα βάλουμε στην άκρη γιατί τα ζήτησε το Συμβούλιο. 21 δι λοιπόν που θα δαπανηθούν το 2019 ανάλογα με τα αποτελέσματα. Οι χώρε που έχουν δαπανίσει τα κονδύλια και μπορούν να δείξουν τα αποτελέσματά του πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδου κονδύλια. Γιατί να περιμένουμε το 2020 φαντάζομαι ότι χώρες που, δεν, χώρες που δεν δαπάνησαν τα κονδύλια και τα έχουν όλα ακόμα στο φάκελο για το 2021-2023. Μπορεί κανείς να σκεφτεί γιατί χρειάζονται αυτές οι χώρες νέα χρήματα, νέους πόρους. Είναι η αρχή μη συν τρία. Ε, και έτσι επενούμε την ε, τεμπελιά. Πρέπει να τα καταδικάζετε αυτό να επιβραβεύουμε τους ε, δραστήριους, αυτούς που πέφτουν με τα μούτρα από την αρχή. Και κλείνοντας, χρειαζόμαστε κάτι σαν θετικό κίνητρο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως ανέφερε ο κύριος Βανιμπρέσκα. Φαντάζομαι οι προτάσεις σας θα προκύψουν από το σύνολο του Σώματος των Επιτρόπων και φαντάζομαι ότι και ο Αντιπρόεδρος θα ασκήσει πιέση για τον εξυγχρονισμό. Οπότε πρέπει να εξυγχρονίσουμε και το εκπαιδευτικό σύστημα όπου αυτό είναι απαραίτητο ή τις ε, δημόσιες προμήθειες. Χωρίς να τα λέμε, τα ξαναλέμε, δέκα χρόνια τα λέμε πρέπει να αναλάβουν και οι κυβερνήσεις τις ευθύνες τους. Και αυτό μπορεί να γίνει στο υψηλότερο επίπεδο της Επιτροπής και του δικού μας. Το ΕΛΚ είναι διαθετημένο να τα συζητήσει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σχεδόν δύο λεπτά πάνω από το όριο βέβαια ήσασταν. Πραγματικά θα πρέπει να επιμείνω στο χρονικό όριο. Ο κύριος Χοφ από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ich äh, Ελπίζω να τηρήσω το χρόνο πως και οι ε, προλαλήσαντες. Ε, θέλω και εγώ να μιλήσω για την εμπειρία. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι μικρή εμπειρία μας. Υπάρχουν πολλά αυτά τα οποία θέλουμε να ε, πετύχουμε και θα πρέπει να σκεφτούμε τι έχει γίνει. Εγώ εκπροσωπώ ένα ε, Λάντα από την πρώην ε, ε, λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας και ακριβώς με την στήριξη των κονδυλίων συνοχής έχουμε πετύχει μεγάλη πρόοδο, αλλά υπάρχουν ακόμη σημαντικές απαιτήσεις και Πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλές αλλαγές ε, τα τελευταία χρόνια και έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις. Έχουμε μεγάλα ζητήματα που αφορούν ε, και που έχουν να κάνουν και με τις δημογραφικές αλλαγές ε, και πραγματικά χρειαζόμαστε κονδύλια της πολιτικής αρχής. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σνάιντερ γιατί έχει αναφερθεί και στην 7η έκθεση αρχής, αλλά για τις ε, ε, τα κρατήδια της ε, τέος ε, λαϊκής δημοκρατίας, κύριε Σνάιντερ, υπάρχει μια παγίδα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά το ίσωμα. Πραγματικά υπάρχουν τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που χρήζουν δικαιολογημένα χρηματοδότησης και υπάρχουν και κάποιες άλλες περιφέρειες που έχουν προβάδισμα εναντίον μας. Μετά το Brexit θα πρέπει να γίνει ένας στατιστικός υπολογισμός. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα και σε αυτό το χάσμα τελικά εμείς και χάσουμε εντελώ ε, τις ε, ε, επιδοτήσεις που παίρνουμε. Τα είπε πολύ καλά ο κύριος Σνάιντερ ότι υπάρχει ο δείκτης του ΑΕΠΑ αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι δείκτες όπως είναι ο δημογραφικός για παράδειγμα. Και ακριβώς επειδή εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή που αντιμετωπίζει σημαντικές εντάσεις, ιδίως δημογραφικές, όταν υπάρχουν πάρα πολλές ε, διαθροτικές αλλαγές, όταν έχουμε την αλλαγή, το μετασχηματισμό της οικονομίας, παροχή υπηρεσιών κτλ. Και έχουμε κάποια χαρακτηριστικά που είναι ιδιαίτερα ε, στις σοσιαλιστικές ε, πρώην, σοσιαλιστικά πρώην κρατή της Γερμανίας. Είναι αισθητά όλα αυτά τα προβλήματα ακόμη και αν μου επιτρέπετε να πω για τα τελευταία δεκατόσα δευτερόλεπτα ότι ναι, ε, άμα μειωθούν τα κονδύλια ε, συνοχής θα πρέπει να υπάρξει ένα πολύ σαφές ε, μια πολύ σαφής διάκριση. Να δούμε γιατί γίνεται αυτό, λόγω των οικονομικών προοπτικών ή για λόγους δημαγωγικούς λαϊκίστικους. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρόνο. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Ντούναη, θα ήθελα να πω, σας ζητώ συγγνώμη αν κάνω κάποιο λάθος με την ακριβή προφορά των ονομάτων. Σας το λέω τώρα γιατί μπορεί να κάνω λάθος ανά πάσα στιγμή. Οπότε σας ζητώ εκ των προτέρων. Συγγνώμη, κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Κυρία Τούνα από το ε, Ουγγρική Εθνοσυνέλευση. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίου, χαίρομαι που παίρνω το λόγο εδώ και που συμμετέχω στη σημερινή συνεδρίαση. Να υπενθυμίσουμε ότι για την Ουγγαρία τα ευρωπαϊκά κονδυλία είναι σημαντικό εργαλείο για την οικονομική και κοινωνική εξίσωση, για την ανάπτυξη και για την διεύρυνση των κοινωνικών ευκαιριών. Στις προηγούμενες περιόδους, χάρη στις χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη, δημιουργήθηκαν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πάνω από 3.900 ερευνητικά προγράμματα υποφελήθηκαν τέτοιων κονδυλίων πολλές εξελίξεις, πολλές υποδομές δημιουργήθηκαν, και διευρύνθηκε και το ευρυζωνικό διαδίκτυο. Πρέπει να επισημάνω ότι στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ε, δύο φορές το χρόνο με πρωτοβουλία της Ουγγαρικής Κυβέρνησης συζητάμε για την ε, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η τελευταία συζήτηση έλαβε χώρο ε, φέτος στις 27 Μαρτίου. Στη συζήτηση αυτή οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων εξέφρασαν τις θέσεις τους σε σχέση με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τώρα, τι γίνεται για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η Ουγγαρία θα ήθελε περισσότερη διαφάνεια και απλούστευση σε θέματα πληρωμών και μηχανισμών. Θεωρούμε επίσης ότι δεν πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση ε, μεταξύ, με το ήπιο σύστημα το να διατηρήσουμε τα, η πολιτική συνοχή σε κάποιο επίπεδο και τη διαδικασία σύγκληση είναι πολύ σημαντικό να μην περιορίσουμε την πρόσβαση στους κανόνες επιλεξιμότητας των κανόνων ε, ε, συνοχής. Επίσης πιστεύω πρέπει να μερεμνήσουμε να, ε, για την θέσπιση κανόνων για την πολιτική συνοχή μετά το 2020 χωρίς να μειωθούν τα κονδύλια για τις χώρες που τα χρειάζονται. Για το νέο προπολογισμό της Ευρώπης και για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε ότι με την αναχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας θα λύνουν 10-12 δισεκατομμύρια από τους πόρους. Οπότε εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι αυτή η μείωση των πόρων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες δυσκολίες που απαιτούν περισσότερους πόρους. Πώς θα επιτύχουμε κάποια ισορροπία. Η επιτυχία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτήθηκε και από την επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Θεωρούμε ότι τα κονδύλια που εκχωρούνται δυνάμει της πολιτικής συνοχής σε περίπτωση που μειωθούν θα οδηγήσουν σε αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά επίσης την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των χωρών και των περιφερειών. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι η Ένωση αποκτά προστιθέμενη αξία από τις επενδύσεις στα κράτη-μέλη και από την ίδια τη συνοχή. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν πρέπει να γίνει σύμβολο αιρεσιμότητας ε, όσον αφορά την καταβολή πληρωμών. Να πω επίση ότι το επίπεδο συγχρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει απαραλλακτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα κάποιον από του σοσιαλιστέ και δημοκράτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Μπρέσο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες τελευταίος ο Γερμανός συνάδελφος που υπενθύμησε πως το θέμα της μελλοντική ε, πολιτικής συνοχής είναι η ανταγωνιστικότητα όλων των περιφερειών. Είναι πολιτική για όλες τις περιφερειές, γιατί όλες οι περιφερειές της Ευρώπης πρέπει σε αυτές τις εποχές κρίσης να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητα που έχουν απολέσει σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Προφανώς ε, διατηρώντας ε, τις διαφορές σε θέματα εσόδων και λαμβάνοντας υπόψη και τις παραμέτρους που προκύπτουν από την εκθέση της Κομισιόν ε, και που αφορούν τα θέματα της ανταγωνιστικής δυσκολίας ε, για διάφορους λόγους δημογραφικούς, επίπεδα παιδείας, ικανότητα καινοτομία, όλα τα ζητήματα, όλες οι παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να μην ε, χρησιμοποιούμε πάντα και μόνο εισοδηματικά κριτήρια. Δεύτερο ζήτημα, η απλούστευση. Αν θέλουμε, ή μάλλον για να συμμετέχουν πραγματικά όλοι οι πολίτες στη διαδικασία που θα οδηγήσει στην αλλαγή της ε, οικονομίας, στην επανεκκίνησή της, για να κάνουμε αυτά λοιπόν θα πρέπει τα προγράμματα που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια να γίνουν πιο κατανοητά για τους πολίτες. Σίγουρα θα υπάρχει ένα πιο τεχνικό κομμάτι το οποίο θα ανταποκρίνεται στι απαιτήσει τη Κομισιόν φυσικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφέ κατανοητό κομμάτι με του μεγάλου στόχου. Όπου θα υπενθυμίζουμε το σύστημα επιχειρήσεων, έρευνα, του πολίτε, ε, ε, όλοι αυτοί οι τομεί θα πρέπει να καταλαβαίνουν τα εγγραφά μα. Αλλιώ δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία τη πολιτική συνοχή. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Πιστεύω ότι για πολλές περιφέρειες, για πολλές περιοχές ε, είναι δύσκολη η προετοιμασία έργων έγκαιρα και να μην χάνουν χρόνο στην υλοποίησή τους όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό κομμάτι των κονδυλίων αυτά που απομένουν ενδεχομένω από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για να προετοιμαστούν για την επόμενη. Και αυτό είναι σημαντικό οι γενικές γραμμές του νέου προγραμματισμού να έχουν καθοριστεί όπως υπενθύμισε η κυρία Κρέλ με τρόπο τέτοιο ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη και στις περιφέρειες να προετοιμαστούν για τη νέα προγραμματική περίοδο και να ξεκινήσουν ήδη από τώρα να προχρηματοδοτούν την ε, προετοιμασία έργων διότι για τα έργα υποδομής ούτως ή άλλως ε, υπάρχει κάποιος χρόνος ε, αρκετά μεγάλος για τα έργα αρχίζει κανεί, δεν αρχίζει κανεί να σχεδιάζει τη στιγμή που λαμβάνει τα κονδύλια, γιατί εκεί έχει ήδη σημειώσει μεγάλη καθυστέρηση για την υλοποίηση. Οπότε, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι απόψει σας. Τι απόψεις των υπευθείων της διαχείριση αυτών των κονδυλίων σε επίπεδο εδαφικό. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω τώρα το λόγο σε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Γάκης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Γάκη, έχετε το λόγο. μικροφώνου είστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ξέρετε, όλοι γνωρίζουν ότι η περιοχή μας, η χώρα μας και ιδιαίτερα η περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, έχει πληγεί από μια πρωτοφανή κακοκαιρία. Με αποτέλεσμα, εκτός από την απώλεια 22 ανθρώπινων ζώων να, και τραυματισμών, να υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή στο σύνολο των υποδομών της πληγή σας αυτής της περιοχής. Γνωρίζουμε τις τεχνικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, Εξαιτία όμω ε, του άκρου επίγοντο και σοβαρού προβλήματο που δημιούργησαν πλημμύρε στην Αττική την προηγούμενη εβδομάδα, ζητάμε την αρρωγή των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τι ελληνικέ υπηρεσίε για την εξέβριση λύσεων μέσω άλλων προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών Ταμείων. Είναι θετικό ότι ε, πρότεινε η κυρία Κρέτσου την απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τέτοιες, για τέτοιες ε, περιπτώσεις. Και είναι επίσης θετικό ότι αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει το πρόβλημα της Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά την, ε, την υπόθεση της προγραμματικής της σύγκλησης, η Ελλάδα υποστηρίζει την ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και την ενδυνάμωση πολιτικών όπως αυτές της συνοχής και της αγροτικής πολιτικής και της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ειδικότερα, η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά, είναι αναγκαία όχι μόνο γιατί έχει συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών και τη μείωση των ανισοτήτων, αλλά και γιατί έχει συμβάλει ουσιαστικά στις ευρύτερες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ευρώπη του 2020. Ωστόσο, η σύνδεσή της με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις ειδικέ αναχώρασεις στάσει θα πρέπει αυστηρά να περιοριστεί σε δεόντως αιτιολογημένες συστάσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση των περιφερειακών ενισχύσεων με την εκπλήρωση των μακροοικονομικών προϋποθέσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά Τη νέα αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής. Μετά το 2020 πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να στηρίζει αναλογικά όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως του επίπεδου, του επίπεδου ανάπτυξης και να μην απευθύνεται μόνο στις λιγότερο αναπτυγμένες, έτσι ώστε να δίνεται δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες να μεγιστοποιούν τις αναπτυξιακές τους ευκαιρίες. Επιπλέον, η μεθοδολογία κατανομής των πόρων της προγραμματικής περίοδου μετά το 2020 θα πρέπει να συμπεριλάβει πέραν του περιφερειακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και άλλους δείκτες οι οποίοι αναδεικνύουν την κοινωνική και χωρική διάσταση της πολιτικής όπως το επίπεδο φτώχειας, την ανεργία, την απασχόληση, την προσβασιμότητα αλλά ε, έτσι ώστε να αποτυπώνεται ακριβέστερα η πραγματική εικόνα των περιφερειών. Εδώ να σημειωθεί το έλλειμμα να μην συμπεριλαμβάνεται στι μετρήσει των περιοχών το άρθρο 174 τη συνθήκη στι νησιωτικέ και ορεινέ περιοχέ. Κάτι που είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση ευνοϊκότερων κατανομών ή και επιλέξιμων για αυτέ τι περιοχέ ε, πολιτική συνοχή. Δράτω την ευκαιρία να αναφέρω και την τροποποίηση του Optimus που συγκεκριμένα στον κανονισμό του ΕΤΠΑ 1301 του 2013 άρθρο 3 το οποίο αφορά έργα πολιτισμού και τουρισμού. Τονίζουμε ότι πρέπει να, αρθεί κάθε περιορισμός προϋπολογισμού στα έργα πολιτισμού και τουρισμού, όπως και στα υπόλοιπα έργα υποδομών που, χρηματοδοτούνται από το, ΕΤΠΑ. Η Ευρώπη, αναγνωρίζοντα τη σημασία του πολιτισμού της, επιβάλλει να τον προστατεύει και να τον αναδεικνύει. Συγγνώμη για το φιαστικό της ε, τοποθέτησή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σμαραντάτσι από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, εμείς χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ρέτζη του Ευρωκοινοβουλίου για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε από κοινού το μέλλον ε, της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί επί μακρόν στις Βρυξέλλες, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι μόνο. Η έκθεση αναλύει την πολιτική συνοχή όσο έχει σήμερα και θεσπίζει ένα πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020. Δεν προδικάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιμένουμε εντός του 2018, όμως ε, τροφοδοτεί τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα και προτείνει μία πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εξυπηρετεί τρεις σκοπούς. Πρώτον, ε, να αξιοποιήσουμε την παγκοσμιοποίηση, να μην αφήσουμε κανέναν εκτός και να στηρίξουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Το ψήφισμα της 13ης ε, ε, Ιουνίου του Ευρωκοινοβουλίου δείχνει ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 και υπογραμμίζει ότι θα ε, πρέπει να υπάρξει συνένεση επί δύο βασικών αρχών μιας πολιτικής συνοχής. Επαρκής προπολογισμό και εξηγέση όλων των περιφερειών και των μεταβατικών και των μη ανεπτυγμένων ε, περιφερειών, στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Η Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, επιθυμούν η μελλοντική πολιτική συνοχή να είναι ευέλικτη, απλουστευμένη και διασυνδεδεμένη. Όλα όσα έχουν υποθεί και γραφεί υπογραμμίζουν ακριβώς την προσθεμένη αξία ε, της πολιτικής συνοχής, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη θα πρέπει να παραμείνει η βασική πηγή επενδύσεων που ε, οδηγεί σε βιώσιμη και ευφυή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες. Όπως ανέφερε και η Επίτροπος Κρέτσου, βρισκόμαστε σε καλή τροχιά σε ό,τι αφορά την πολιτική συνεχής μέχρι το, συνοχής μέχρι το 2020. Το μέλλον της πολιτικής συνοχής πάει χέρι-χέρι με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σύγχρονη, ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχή που να οδηγεί σε ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλε τι περιφέρειε. Το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 θα πρέπει να δίνει όλα τα μέσα στα κράτη-μέλη για να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχή, η οποία θα πρέπει να διδραματίσει κεντρικό ρόλο ε, στο, στη μελλοντική διαμόρφωση του υπερπολογισμού. Είναι η μοναδική πολιτική που απευθύνεται σε όλα τα κράτη-μέλη και τους επιτρέπει να σημειώνουν πρόοδο σε τομείς κλειδιά για την Ευρώπη. Η περιφερειακή πολιτική έχει πραγματική προσταθεμένη αξία και αυτό φαίνεται και από την 7η έκθεση για τη συνοχή. Αποδεικνύει ότι η πολιτική συμβάλλει στη σύγκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούμε ότι στην πολιτική συνοχή θα πρέπει να αυξήσουμε τη σημασία της ε, εδαφικής προσέγγισης και της ολοκληρωμένης ε, διαχείρισης. Γιατί σε αυτό το επίπεδο είναι που έχουμε την καλύτερη αξιοποίηση. Και τελικά αυτές οι επιχειρήσεις δείχνουν ε, απτά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να ταυτοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο απλούστευσης της πολιτικής συνοχής και έτσι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων και να πετύχουμε ε, συγκεκριμένους στόχους που θα είναι επωφελείς και για τους δικαιούχους και για τις ε, αρχές διαχείρισης. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της σταθερότητας μέσω και μακροπρόθεσμα, όπως αναφέρεται και στο προγραμματικό έγγραφο. Χρειαζόμαστε περισσότερο στονισμό και ε, μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμβάλλουμε όσο μπορούμε καλύτερα στη διαμόρφωση αυτή τη πολιτική. Πρέπει η πολιτική συνοχή να διατηρήσει έναν κέριο ρόλο στο ε, επερχόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και παραμένουμε στη διάθεσή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Είπα ότι θα επιμείνω ε, στο χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε τώρα με την κυρία Μιχέλς. Παρακαλώ. Μιχέλς, Μισελς. Μίχελς. Ευχαριστώ πολύ. Πολιτική συνοχής. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της αλληλεγγύης. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό νομίζω. Νομίζω ότι λίγο πολύ συμφωνούμε όλοι από αυτού. Μάλλον Περισσότερο παρά λιγότερο, συμφωνούμε. Αλλά θα πρέπει να μην βγούμε από αυτή την αίθουσα με μια αισιοδοξία υπερβολική ότι τα έχουμε πετύχει όλα. Και πραγματικά υπάρχουν εκτός ε, της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης και εκτός ε, του Κοινοβουλίου άλλες τάσεις και άλλες επιθυμίες και υπάρχουν και άλλες στρατηγικές όπου δεν περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής. Υπάρχει η τάση να κάνεις λιγότερα, ε, με λιγότερα χρήματα περισσότερα πράγματα. Υπάρχει και αυτή η τάση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε πάντο δυνατόν ώστε μαζί όλοι τα εθνικά κοινοβούλια και σε όλα τα επίπεδα επίπεδο ευρωπαϊκό, εθνικό, επίπεδο κρατηδίων, περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες και να διακηρύξουμε την ανάγκη για την ε, συνέχιση πολιτικής συνοχής. Θέλω να πω ε, ποια είναι η δική μας θέση. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι περιφέρειες ε, ε, θα πρέπει να μπορούν ε, να παραμείνουν επιλέξιμες. Από την Θουριγκία μίλησε ένας ε, Γερμανός συνάδελφος και περιέγραψε την κατάσταση των κρατηδίων της Τέος Ανατολικής Γερμανίας. Πραγματικά σίγουρα δεν θα πρέπει να υπερεπεξεργαστούμε την νομοθεσία. Πρέπει να απλουστευτεί και πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία αλλά ε, πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι που το συζητούμε εδώ και χρόνια. Αλλά συγκεκριμένες προτάσεις ακόμη δεν υπάρχουν επιτάπητος. Εμείς λοιπόν θεωρούμε και θέλω να το πω ξεκάθαρα αυτό ε, ως ενωμένη αριστερά ε, στο Κοινοβούλιο εμείς παραμένουμε και επιμένουμε ε, για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Πρέπει να καταργηθεί κατά την άποψή μας. Επίσης πρέπει να γίνει μια διακήρυξη, μια δήλωση προθέσεων. Ακούμε και από την Κομισιόν και από άλλους πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά, αλλά το μέτρο ε, και ο πύχης ε, για την πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους κάποια στιγμή να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι και να πάψουν πλέον μόνο οι δηλώσεις και οι διακηρύξεις ε, που δεν έχουν περιεχόμενο. Μόνο τότε μπορούμε να συζητήσουμε πραγματικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Λούτβικ από το γερμανικό Bundestag. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, είμαι από το Βραδεμβούργο και την οικονομική μας ε, άνοδο την ε, χρωστάμε ε, στα ταμεία και τα κονδύλια συνοχής. Ήμασταν, ε, όταν ξεκίνησε η περιοχή μας ήταν ε, από τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τώρα είμαστε από τις πλέον ανεπτυγμένες ε, και άρα έχουμε ιδέα εμπειρία. Και μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί η πολιτική συνοχής. Βλέπει κανείς τις επιτυχίες και πραγματικά έχει αποτελέσματα η πολιτική συνοχή. Ε, βέβαια υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μια τελμάτωση στην οικονομική ανάπτυξη. Βλέπουμε να προελάβουν τα εθνικιστικά κινήματα, τα λαϊκιστικά κινήματα και πραγματικά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και ισχύ στην πολιτική συνοχή ε, γιατί ε, θα βοηθήσει πάρα πολύ και η εξάλληψη των ανισοτήτων. Βέβαια ε, και οι ευρωπαϊκοί στόχοι και προτεραιότητες θα πραγματοποιηθούν μόνο αν οι περιφέρειες είναι μαζί, αν συνδέονται στις προσπάθειες. Και θα πρέπει επίσης πολιτική συνοχή και τα αποτελέσματά της να είναι ορατά επιτόπου. Και πρέπει να πετύχουμε αυτούς τους στόχους για να έχουμε μια κοινή ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και την ευρωπαϊκή αυτή προστέμενη αξία θα πρέπει να την κάνουμε ορατή. Γιατί πραγματικά ε, υπάρχει και το ζήτημα της επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς προβάλλουμε τα επιτεύγματά μας. Μετά το 2020 θα πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες και οι πολιτική συνοχή να έχει έναν προεξάρχοντα ρόλο. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη απλούστευση. Αν θέλουμε να είναι και πιο ορατή η πολιτική συνοχή, θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει διοικητικό άχθος, γραφειοκρατικό άχθος, το οποίο είναι πάρα πολύ ορατό. Και αυτό αφορά όχι μόνο την πολιτική συνοχή, αλλά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. πρόταση ε, είναι πολύ θετική, αντί να έχουμε μια ριζική ε, αναδιάρθρωση, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του τοπικού επίπεδου πλέον και επίσης να υπάρξει και μεγαλύτερη καταπολέμηση της διαφθοράς και των απατών. Δεν μιλάω βέβαια για μια ε, επανακρατικοποίηση τη πολιτική συνοχή. Φυσικά οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητε ε, τη περίοδου προγραμματισμού θα τίθεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ε, διοικητικά και τεχνικά νομίζω ότι εμεί μπορούμε σε τοπικό επίπεδο να εφαρμόσουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γνωρίζουμε και εδώ και δεκαετίε ε, ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε τι πολιτικέ συνοχή. Και Σίγουρα καλό είναι να υπάρξουν και κάποιες διαφοροποιημένες ε, προσεγγίσεις. και θα πρέπει σίγουρα ε, να ληφθεί πολύ περισσότερη υπόψη η αρχή της αναλογικότητας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βόησετσόφσκι, αν το λέω σωστά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή. Έρχομαι από την Πολωνία. Είμαι αντιπρόεδρος μιας ε, τοπικής αρχής. Στο μέλλον της πολιτικής ε, συνοχής θα πρέπει να μας αποσχολήσει περισσότερο η ύπεθρος. Η έκθεση δείχνει ότι έχουμε χάσει περίπου 4 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Από τα 14,5 πήγαμε στα 7 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι χάνουμε χίλιους γεωργούς κάθε χρόνο. Επίσης, βλέπουμε ότι Αυξάνεται και η μέση ηλικία των γεωργών. Πλέον περισσότεροι είναι άνω των 45 ετών. Αν διαβάσετε τα έγγραφα του Ελληνικού συνεδρίου, υπάρχουν περιοχές όπου το 40% των γεωργών είναι άνω των 60 ετών και σε ορισμένε χώρες ακόμα περισσότερο. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Ενδεχομένως λοιπόν να χάσουμε τη γεωργία στην Ευρώπη και έτσι και την επιστηστική μας ασφάλεια. Η κοινή γεωργική πολιτική δεν φτάνει για να κρατήσει τους γεωργούς ε, στην Ήπεθρο και για να ε, αποτρέψει ή να αναστρέψει ε, τη γύρανση του πληθυσμού. Πρέπει να διασφαλίσουμε περισσότερη στήριξη προς τη γεωργία, αντλώντας πόρου από την πολιτική συνοχή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει περισσότερη πρόσβαση ε, στο, στην περίθαλψη, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην Πολωνία. Αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα με τα σχολεία ε, στην Ήπεθρο. Οι μαθητέ πρέπει να βγαίνουν ε, μεγάλε αποστάσει για να φτάσουν στο σχολείο και ίσω αυτό να είναι και μία από τι βασικέ αιτίε που κάνουν τον κόσμο να φεύγει από την Ήπεθρο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική που είναι απαραίτητη ε, δεν μπορεί από μόνη της να κρατήσει τους γεωργούς στην Ήπεθρο. Πάνω από το 90% της επικράτειας ε, αφορά τον γεωργικό κλάδο στη χώρα μου. Αλλά έχουμε δώσει μόνο 10% των κονδυλίων από την πολιτική συνοχής. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει ε, να σκεφτούμε περισσότερο τον γεωργό στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βάνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή αυτή απόψεων με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβουλία χθε ε, είδα ε, κάποιους ε, επικεφαλής πολιτικών ομάδων που είχα μια συνεργασία και με, συνάντηση με τον κύριο Ταγιάννη. Ήταν εκεί και από την Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση κάποιοι συνάδελφοι. Συζητήσαμε λοιπόν με την βουλγαρική πλευρά και νομίζω ότι πραγματικά με πολύ θετικό, σε πολύ θετικό κλίμα συζητήσαμε όλα αυτά τα στήματα, τις διαφορές, μιλήσαμε για την ανάγκη ενδυνάμωση ενδυνάμωσης της πολιτικής συνοχής και ακριβώς ε, τις προβλεπόμενες περικοπές. Ε, όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ξέρετε ότι ε, μετά την Εστονία έπεται ε, η Αυστρία και η Ρουμανία και η Βουλγαρία βέβαια. Και όλα αυτά τα συζητούμε γιατί η πολιτική συνοχή ε, τώρα μόλις ξεκινάει να τελεί πραγματικά αντικείμενο συζήτηση ε, και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε παραπάνω από έτοιμοι και διατεθειμένοι να βρούμε τις λύσεις για την πολιτική συνοχή πριν τις επόμενες ευρωεκλογές. Ε, πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πολιτική συνοχή. Σε αυτό το βλέπουμε με τα αποτελέσματα επιτόπου, κυρίως ε, για την εδαφική ε, συνοχή και την κοινωνική την οικονομική. Θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, την ανεργία και να στηρίξουμε ε, τις πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα των τάμιων και βέβαια και την κλιματική αλλαγή να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα υπάρχει το ζήτημα της διαμόρφωσης της ε, πολιτικής συνοχής ε, και της πρικοδότησης της, δηλαδή ποια είναι τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα. Πραγματικά ε, θα τα δούμε όλα αυτά πάρα πολύ προσεκτικά. Υπάρχει και η κριτική του ελεγκτικού συνεδρίου για το υπόσχεσμο τα κονδύλια. Έχουμε το ΕΦΣΙ, δηλαδή το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker ε, και αυτό δεν πρέπει να το δούμε ως πανάκια το εύση γιατί δεν μπορεί να ε, εξουδετερώσει και να παλείψει τις διαφορές και τις ανισότητες μεταξύ ε, περιφερειών. Μόνο το 4% ε, των ε, κονδυλίων από το σχέδιο Γιούνκερ πηγαίνουν στις κοινωνικές υποδομές και αυτό είναι κάτι πραγματικά ελάχιστο για την, ε, το μέλλον τώρα της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ πιο στενή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Είμαι πεπισμένη ότι μακροπρόθεσμα έτσι θα μπορούμε να βρούμε πιο βιώσιμες λύσεις για τους ε, συμπολίτες μας. Το που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση και συμφωνώ με την προλαλή σας Ευρωβουλευτή φυσικά και δεν θέλουμε η πολιτική συνοχή ουσιαστικά να είναι ένα τιμωρητικό μέσο ε, να τιμωρεί ε, τις περιφέρειες. Αν έχουν δηλαδή ληφθεί λάθος αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο να χρεώνονται τα λάθη αυτά οι περιφέρειες. αφορά δηλαδή και τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, ε, τα κριτήρια ελλείμματος ε, και να οδηγεί η παραβίαση εντό εισαγωγικών κάποιων όρων, το είδαμε με την Πορτογαλία, το είδαμε με την Ισπανία, να περικόπτονται οι πόροι. Σίγουρα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη πιο πολύ τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου. αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητα και γι' αυτό θα πρέπει ε, να δούμε και τα σχετικά με τη διαδικασία του ΑΤΡΕΠΤΑ. 7. Υπό αυτό το πρίσμα δεν θα πρέπει λοιπόν να εστιάζουμε μονόπλευρα ε, στο ΑΕΠ ως δίκτυ για την κατανομή των πόρων, ε, το καθάριστο ε, προϊόν, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλα κριτήρια αναπτυξιακά, κοινωνικά, δημογραφικά και άλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η κυρία Ντένσκι από το Δανέζικο Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω ότι γενικά τόσες πολλές χώρες ε, εποφελούνται από την πολιτική συνοχής. Και εμείς έχουμε επωφεληθεί σε ορισμένους τομείς στη Δανία. Αλλά πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Υπάρχει μια παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη οπωσδήποτε. Και αυτή είναι είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου των περιοχών που υποφέρουν από την αστικοποίηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανεξαρτήτως το αν μια χώρα είναι πλούσια ή φτωχή, οι προκλήσεις είναι οι ίδιες. Και αν τα κονδύλια δίδονται μόνο στις φτωχές χώρες, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στις πλούσιες και αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε από αυτή την πτυχή την πολιτική συνοχής. Όσον αφορά το ευρυζωνικά δίκτυα, δεν ξέρω στις δικές σας ε, χώρες, αλλά στη Δανία έχουμε καθήκον να παρέχουμε νερό, ηλεκτρισμό και θέρμανση και σταθερές τηλεφωνικές γραμμές ε, σε όλους. Ε, πρέπει να το όλοι υποχρεούνται να το παρέχουν αυτό, αλλά σήμερα έχουμε και την υποχρέωση να παρέχουμε ευρυζωνικό δίκτυο. Αλλά είναι, γιατί είναι δύσκολο να πληρώσει κανεί του λογαριασμού του χωρί διαδικτύο ή να διαβάσει τα διάφορε ανακοινώσει του δημόσιου τομέα. Ε, και πολλέ ειδοποιήσει του δημόσιου τομέα έρχονται μέσω διαδικτύου και δεν έρχονται με, την με το κανονικό ταχυδρομείο, οπότε υπάρχει αυτή η υποχρέωση να παρέχουμε ευρυζωνικά δίκτυα σήμερα. Επίσης μιλήσαμε για τις θέσεις εργασίας. Στις αγροτικές περιοχές, δυστυχώς, Ο κόσμος επίσης υποφέρει από την αστικοποίηση, διότι οι δουλειές έχουν μεταφερθεί στα αστικά κέντρα. Για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σε αυτές τις περιοχές πρέπει να κάνουμε κάτι. Στη Δανία 4.000 θέσεις εργασίας ε, ε, του δημόσιου τομέα μεταφέρθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Ε, αποτελούν πλεονέκτημα για αυτές τις περιοχές διότι σε μια περιοχή όπου υπάρχουν 200 δουλειές θα ανοίξει και ένα καφέ, ένα κομμωτήριο, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και αυτό θα σημαίνει ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν θέσει εργασία. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στην κυρία Ντεμάτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, εθνικοί και ευρωπαίοι, είναι κακή η πολιτική συνοχή ε, να σας ζητήσω να μιλάτε πιο κοντά εθνικοί βουλευτές και συνάδελφοι εδώ του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι λόγω της κακής ε, αντίληψης της πολιτικής συνοχής ε, ε, οι πολίτες μας είναι δύσπιστοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνουν το στόχο της συνοχής, δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες ούτε τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, στη δική μου εκλογική περιφέρεια στο νότο της Ιταλίας, λόγω της έλλειπους πληροφόρησης αλλά και επειδή η χρήση των κονδυλίων είναι αμφίβολη, για να το πω έτσι, δεν είναι πιστευτή αυτή η πολιτική. Ε, για παράδειγμα, χρηματοδοτούν πράγματα περίεργα. Ε, υποτίθεται ότι δημιουργούνται θέσει εργασία ε, και χρησιμοποιούνται ξαφνικά 2.000 ημέρες για να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση. Ή ε, χρειάζονται δύο χρόνια για να εγκριθεί ένα έργο για να αφήσουμε στο πλάι τη χρήση των κονδυλίων που είναι αμφίβολη και τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Όπως φαίνεται όμως η πρόταση αυτής της Επιτροπής θα είναι μια μεταρρύθμιση που θα υφίσταται περισσότερο σε προϋποθέσεις, δημοσιονομικές δεσμεύσεις και ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ απευθύνομαι τώρα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Πώς εξηγείτε ε, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις περικοπές ε, των συντάξεων, ε, και ότι παρόλα αυτά δεν θα υπάρχουν πλέον ευρωπαϊκά κονδύλια να ξοδευτούν. Ε, αυτή είναι η μόνη πολιτική που κατανέμει πόρους πραγματικά, αλλά δεν το κάνει σωστά. Δεν έχει νόημα να λέμε συνέχεια πόσο αναγκαίες είναι οι επενδυτικές πολιτικές. Κάνω έκκληση στις κυβερνήσεις, ειδικότερα στη δική μου στις πολιτικές δυνάμεις, που την υποστηρίζουν στο Δημοκρατικό Κόμμα και στο κεντροαριστερά. Ε, σταματήστε να περικόπτετε ε, τα χρήματα για τις φτωχές περιοχές. Σταματήστε να έχετε τον αποκλεισμό αυτών των περιοχών. Αγωνιστείτε ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιηθεί για ένα ελάχιστο εισόδημα που δεν υπάρχει ούτε στην Ιταλία ούτε στην Ελλάδα. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, τι κάνετε για αυτή τη μάχη, το ΕΛΚΑ και το Φόρτσα Ιτάλια εκτελείται πιστά οτιδήποτε σας λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Από την Επιτροπή ΡΕΤΖΙ, τα μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν, κυρία Μόλκοβα. Σμόλκοβα, μάλλον έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω για ένα ζήτημα για το οποίο δεν μιλήσαμε ακόμα αφού μιλάμε για πολιτική συνοχή. Ένα ζήτημα που με απασχολεί, οπότε θα ήθελα να το αναφέρω και σε αυτή τη συνεδρίαση. Σίγουρα δεν έχουν όλοι την πληροφορία αυτή. Θα ξέρατε ότι τον Οκτώβριο, ε, που μόλις πέρασε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εγκρίθηκε ο κανονισμός του Δουβλίνου. Πολύ περιπλοκός. Ήταν πολύ περιπλοκή διαδικασία η έγκριση. Συμφωνώ και εγώ στο ότι ήταν αναγκαίο να εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, αλλά υπάρχει μια τροπολογία που δεν έχω καταλάβει. Ένα άρθρο μάλλον που δεν έχω καταλάβει. Σε αυτό το άρθρο λέγεται ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις ε, υπό τη μορφή μειώσεων κονδυλίων στα κράτη-μέλη που δεν σέβονται το σύστημα μετεγκατάστασης των προσφύγων μεταναστών. Δεν καταλαβαίνω πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί αυτό το, ε, αυτή η αρχή οι μεταναστές δεν θα υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν ακόμα και το 2020. Εγώ είμαι υπέρ της αλληλεγγύης, είμαι υπέρ του γεγονότος ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν από κοινού στην κοινή πολιτική ασύλου και να μοιράζονται και τις ευθύνες και η ιδέα όμως της μείωσης των κονδυλίων σε περίπτωση που δεν δεχθούν πρόσφυγες μου κάνει αλλά όταν επιβάλλουμε κύριο στα κράτη και όχι στις περιφέρειες θα πρέπει να ε, επιβάλλουμε κυρώσει στα κράτη και όχι στι περιφέρειε, γιατί συνήθω δεν είναι λάθο των περιφερειών όταν τηρείται αυτή η, η πολιτική. Τα κράτη αποφασίζουν τέτοια συμπεριφορά. Οπότε ήθελα να ε, αξιοποιήσω την ευκαιρία που είμαι εδώ για να κάνω έκκληση στου εκπροσώπου του Συμβουλίου και τη Κομισιόν και ελπίζω να μα δώσουν μια απάντηση σύντομα σε αυτό το ερώτημα. Εσεί πώ το βλέπετε, πώ φαντάζεστε ότι θα διαχειριστούμε στο μέλλον αυτό το θέμα, γιατί μετά το Brexit θα έχουμε λιγότερα κονδύλια και το, να τα μειώσουμε ακόμα περισσότερο λόγω λανθασμένων αποφάσεων κάποιων κρατών μελών για τις πιο φτωχές περιοχές θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά. Ευχαριστούμε κύριος Παπαδημούλης, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μέσα σε αυτή την αίθουσα η μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ των πολιτικών συνοχής. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο ούτε στην Κομισιόν, ούτε στο Συμβούλιο, εκεί που θα παρθούν οι αποφάσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 2020 και μετά. Πριν δύο εβδομάδες ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, μας είπε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ότι στα χρόνια της κρίσης αυξήθηκαν οι ανισότητες και οι κοινωνικές και οι περιφερειακές. Επομένως, αν θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτή την αύξηση των ανισοτήτων η πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχυθεί και όχι να την αντιμετωπίσουμε ως business as usual. Και δυστυχώς, κύρια Πρόεδρε, υπάρχουν ορισμένοι που έχουν χειρότερα σχέδια από το business as usual. Θέλουν να μειωθούν τα κονδύλια για την πολιτική συνοχής. Γιατί για να έχουμε πολιτική συνοχής ισχυρή χρειαζόμαστε και απλούστευση, συμφωνώ με τον Γερμανό συνάδελφο, αλλά χρειαζόμαστε και πόρους και οι πόροι αυτοί, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνοχή, πρέπει να πηγαίνουν περισσότερο εκεί που υπάρχει ανάγκη. Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια, μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη αποεπένδυση, γιατί αλλιώς δεν υπηρετούμε την πολιτική συνοχής. Θέλω να σας πω πολύ καθαρά τη γνώμη μου. Η κυρία Κρέτσου, η Επίτροπος Κρέτσου, είναι υπέρ της πολιτικής συνοχής αλλά μέσα στην Κομισιόν υπάρχει και ένα στρατόπεδο που προσπαθεί να αποδυναμώνει την πολιτική συνοχή. Και θα ήθελα να ακούσω τι λέει για την πολιτική συνοχή και ο αρμόδιος επίτροπος για τον προϋπολογισμό, ο κύριος Έτιγκερ. Γιατί δεν τον βλέπω να υποστηρίζει τόσο πολύ την πολιτική συνοχή. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει από αυτήν εδώ την αίθουσα, από την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, από τους εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, και χαίρομαι που συμφωνεί και ο συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο Βανίστερ Ρόι, να υπάρχει μια ισχυρή πίεση να μην είναι η πολιτική συνοχής το θύμα του Brexit και το θύμα των περικοπών στον προϋπολογισμό. Και συμφωνώ και με την κυρία Κρέλ που είπε επιτέλους ας φύγει αυτό το παράλογο αίτημα του άρθρου 23 για την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα γιατί έτσι με αυτό το δόγμα τιμωρούνται οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτά τα χρήματα, όπως σωστά είπαν και οι συνάδελφος από τη Ρουμανία και οι συνάδελφος από τη Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γρήγορα να σας απαντήσω ότι αύριο θα έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε τον Επίτροπο Έντιγκερ ό,τι θέλετε και όλη η Επιτροπή θα ακούσει τι απαντήσει. Η κυρία Ροντρίγκε, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώ ε, προερχόμαστε και από αυτόνομη περιφέρεια. Ε, εξαρτώμεθα πλήρω από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Περιμένουμε ακόμα ε, την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που ακούω περισσότερες φωνές υπέρ της ε, κατάργησης του άρθρου 23, γιατί είναι κάτι το οποίο υποσκάπτει την ε, πολιτική συνοχή. Ήθελα να αναφερθώ στα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με το πνεύμα της ε, πολιτικής συνοχής. πάντα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη παραδοσιακά εκφράζεται με επιδοτήσεις ε, προς αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία λοιπόν ε, κάποιες φορές είναι χρήσιμα, άλλες ε, λειτουργούν τιμωρητικά και το Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει θέση ως προς αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι το μέλλον της πολιτικής συνοχής δεν είναι μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων. Ακούω με μεγάλη χαρά τον εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο να λέει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη εκτέλεση των κονδυλίων προ τα κράτη-μέλη. Αυτό όμω τι σημαίνει και ότι θα υπάρξει σημαντική απλούστευση. Τι σημαίνει όμως αυτή η απλούστευση. Δεν με απασχολεί που χρησιμοποιείτε τον όρο ε, απλούστευση, αλλά γιατί μιλάτε για ριζική απλούστευση, radical. Πώ ακριβώς θα παρακολουθείτε αυτή η διαχείριση, Ποιο θα είναι ο ρόλος ε, των ε, διαχειριστικών φορέων πρέπει ο κάθε φορέας να έχει ξεκάθαρη αποστολή, ξεκάθαρη αρμοδιότητα μετά το 2020 και για μένα το μέλλον της πολιτικής συνοχής καθώς και το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τη δυνατότητά μας να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες δεν θα χάσουν την πίστη τους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να καλωσορίσω συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους προσκεκλημένους. Ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, θα θέλω να τονίσω τη σημασία της σημερινής συνάντησης για την πολιτική συνοχή σε μια χρονική στιγμή που όπως είδαμε Ε, βλέπουμε ότι και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν τα, ο καθένα τα έγγραφά του και τι προτάσει του. Η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πολύ ε, σημαντική. Είναι σημαντικό ο ρόλο των κρατών μελών και του Συμβουλίου, όχι μόνο για την διασφάλιση τη επικουρικότητα, αλλά και σε τέτοιου είδου ε, διακοινοβουλευτικέ συνεδριάσει ε, προκειμένου να είμαστε όλοι καλά ενημερωμένοι, προετοιμασμένοι και να λειτουργούμε ε, με δημοκρατικό πνεύμα. Θα ήθελα να επισημάνω και τον ε, κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια στα όσα ανέφερε και η Επίτροπος Κρέτσου και η Κόνσταντς Κρέλ, δηλαδή την έλλειψη προβολής των ωφελών ε, της πολιτικής συνοχής. Και νομίζω ότι ε, την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Επιπλέον, θεωρώ ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν περιφέρειες που σημαίνει ότι οι χώρες είναι δικαιούχοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι περιφέρειες τελικά είναι δικαιούχοι των κονδυλίων. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αποτελέσει και στο μέλλον το βασικό επενδυτικό εργαλείο για την Ένωση. Δεδομένη τη ε, εδαφική, οικονομική και κοινωνική διάσταση. Και όλα αυτά εγγράφονται και στι συνθήκε. Πρέπει ε, λοιπόν ο μηχανισμό να απλουστευτεί, να βασίζεται στα αποτελέσματα και τα κριτήρια παρακολούθηση θα πρέπει να υφίστανται, αλλά με απλούστερη μορφή. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον. Γιατί θα πρέπει να επιτρέψουμε, επιστρέψουμε αρμοδιότητες και στο τοπικό επίπεδο. Κύριος Τζέλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε σε ό,τι αφορά τα διαθετικά ταμεία. Πραγματικά είναι ίσως το σημαντικότερο επενδυτικό μέσο και θα πρέπει να παραμείνει για τις ε, περιφέρειες. Βέβαια, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, φοβούμεθα ότι ουσιαστικά ε, είναι καταδικασμένο σε θάνατο αυτό το πολύ αποτυχημένο κατά το παρελθόν εργαλείο. Σε ό,τι αφορά την απαλλαγή του 2015, είδαμε ότι με τη νέα περίοδο ε, προγραμματισμού ε, δεν ε, είχαμε κάποια θετική, δεν αναφέρθηκε μάλλον κάποιο κράτος και το ίδιο και το 2016. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης Πράγματι υπάρχουν προβλήματα με την ε, νέα περίοδο προγραμματισμού για πολλά, ε, πολλές ε, περιοχές που δικαιούνταν, ήταν δικαιούχοι, ήταν επιλέξιμες περιφέρειες για, τα κονδύλια και θα τα χάσουν αυτά τα δικαιώματα. Επίσης έχουμε παρατηρήσει πολύ μεγάλη δαπάνη. ξέρω έναν σε ένα γραφείο διαχειριστικό και μου είπε πόσες διαδικασίες, ε, ε, πόσες υπογραφές έπρεπε να συλλέξει, ενώ μπορεί να ξεκίναγε από 100, ε, μετά έγιναν 2.000 στην επόμενη, στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού και τώρα έχουν φτάσει σχεδόν στις 2.000. Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να αναλάβουν ε, την εκτέλεση επιτόπου. Ε, υπάρχει και το οικονομικό επιτελείο, υπάρχουν ε, αυτοί οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν, γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν όλοι μαζί και να το λύσουν συλλογικά το πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές ασφάλματα Είναι πολύ σημαντικό με τους συναδέλφους ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια να καθόμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά. Σίγουρα εκεί πονάει πιο πολύ ο λεγόμενος ε, κανονιστικός υπερθεματισμός και υπάρχουν ε, πάρα πολλά νέα ε, νομοθετήματα τα οποία πρέπει και προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται. Όπως σας είπα, από 200 μπορεί να είναι 2.000 οι προδιαγραφές αυτές και δυσκολεύεται πάρα πολύ το έργο των διχειριστικών φορέων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, υπάρξει απλούστευση και επίσης ε, έτσι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά στις περιφέρειες τα επιχειρησιακά προγράμματα. Αλλιώς θα έχουμε καθυστερήσεις ε, όπως αυτές που διαπιστώνουμε σήμερα. Και επαναλαμβάνω το μέλλον των διευθυντικών ταμείων ε, και του Ταμείου ε, Συνοχής είναι πραγματικά σε κίνδυνο. Μιλήσατε για τους φίλους της συνοχής, πράγματα. Σχεδόν από τα στόματα όλων των επιτρόπων μέχρι πριν από κάποια χρόνια άκουγα πόσο σημαντικό, το σημαντικότερο μάλιστα λέγανε είναι το ε, κονδύλι, το, Ταμείο Συνοχής ως εργαλείο για τη δημιουργία νέων θέσεων Δεν ακούω τίποτα πλέον. Το είπε και η κυρία ε, Μίχελς ε, ότι δεν αναφέρονται πλέον αυτά ακόμα και στα έγγραφα της Κομισιόν. Πρέπει επίσης να δούμε το θέμα της... Ε, συγκέντρωσης ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης λέγεται το Ταμείο, άρα δεν μπορεί να γίνονται και να αποφασίζονται όλα κεντρικά. Θα πρέπει ε, να υπάρχει ε, η δυνατότητα να μην προωθούν τα κράτη τις εθνικές τους ατζέντε, αλλά περιφερειακά και τοπικά να γίνεται δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή αποτελεί την βασική, ε, το βασικό θεμέλιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό είναι αναμφίβολο. Αυτό που είναι κρίμα είναι ότι εκφράζονται τόσο πολλές αμφιβολίες τώρα που η πολιτική αυτή ακριβώς αρχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο τις ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σνάιντερ ήθελα να πω αυτό που είπε. Όσο περισσότερε αρμοδιότητε πρέπει να δώσουμε περισσότερε αρμοδιότητες και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις περιφέρειες. Αυτό θα αποτελέσει το κλειδί για την πολιτική συνοχή. Ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, να είναι πιο σαφής, ώστε να λάβει τέτοιε διαστάσεις που να μην τις συζητάμε μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οι αποφάσεις ε, να λαμβάνονται σιγά σιγά και από τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές γιατί αυτές γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζονται. Σήμερα υπάρχει μεγάλο χάσμα όχι μόνο μεταξύ περιφερειών αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές ε, περιφέρειες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν προβλήματα ενότητας στο εσωτερικό τους, είδε. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο την πολιτική συνοχής. Ωστόσο, αυτό θα απαιτήσει μεγαλύτερη ευελιξία, πιο ευέλικτη προσέγγιση και να δώσουμε τη δυνατότητα στις περιφερειακές αρχές να λαμβάνουν αποφάσεις. Πρέπει να τους δώσουμε περισσότερη, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις περιφερειακές ε, αρχές ώστε να έχουμε κάποια προστιθεμένη αξία για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας καλώ να έρθετε στην Πολωνία για να δείτε. Έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Μπόγκοβιτς. Καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι εδώ είμαστε φίλοι της πολιτικής συνοχής και υποστηρίζουμε την αρχή της αλληλεγγύης ε, στην οποία βασίζεται. Η πολιτική συνοχής ε, είναι η κόλλα που κρατά ενωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών ε, εξακολουθούν να υπάρχουν και θα χρειαστεί να βρούμε απαντήσεις και για το μέλλον. Όλοι συμφωνούμε ότι σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλου αριθμού προκλήσεων στην Ευρώπη. Το Brexit, ε, τη μετανάστευση. Θα χρειαστεί να κατανομηθούν ε, κονδύλια ε, για να αντιμετωπιστούν άλλα προβλήματα όπως είναι κατανοητό. Από την άλλη ε, χάνουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι ε, σημαντικός συμμετέχων οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για την κατανομή του βάρους στα άλλα κράτη-μέλη. Τώρα όσον αφορά τα Εθνικά Κοινοβουλία θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα συζητήσετε αυτά και στις χώρες σας και όταν έρχονται οι πρόσωποι σα στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάνε στι Βρυξέλλε λέγοντα το ίδιο που λένε και στι χώρε του. Αλλιώ ε, η πολιτική συνοχή θα αντιμετωπίσει σημαντικέ δυσκολίε. Εμεί οι ίδιοι είμαστε αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτή τη ε, πολιτική ε, συνοχή. Είναι πράγματι οι κανόνε τόσο περίπλοκοι, σίγουρα. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε και γιατί οι εθνικές δομές χρειάζονται τόσο πολύ χρόνο για να υλοποιήσουν την πολιτική συνοχή και τα σχετικά κονδύλια. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υλοποιήσουμε ε, την προοπτική 2014-2020 διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Εγώ ίδιος έχω υπάρξει ε, υπουργό επιφορτισμένος με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Υπέθρου. Ήμουν αρμόδιος για τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Είχαμε συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και στις πρωτεύουσέ μας. Το έχουμε ήδη συζητήσει επαρκώς σήμερα. Θα πρέπει να προβάλλουμε και περισσότερο την πολιτική συνοχής, να γίνει πιο γνωστή. Οι πολίτες μας θα πρέπει να καταλάβουν τη χρησιμότητα της πολιτικής συνοχής, ότι καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο όμορφη, πιο αποτελεσματική, πιο σημαντική. Ευχαριστούμε και τελευταία ομιλήτρια από την Επιτροπή Ρέτζη, κυρία Μάλαντιτς. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων και χαρούμενη που έχουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας το μέλλον της πολιτικής συνοχής και την 7η έκθεση συνοχή. Τρία μηνύματα θα ήθελα να αποστείλω. Πρώτον, αν θέλουμε ισχυρή Ευρώπη, χρειαζόμαστε περισσότερη συνοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο προπολογισμό ε, ε, για τη συνοχή στο επόμενο ΠΔΠ δεν μπορεί να μειωθεί. Είτε να μείνει ο ίδιο, είτε να αυξηθεί. Δεύτερο μήνυμα για την γραμμή προπολογισμού τη Ευρωζώνη. Δεν γίνεται ε, να έχουμε αυτή την γραμμή προπολογισμού σε βάρο τη πολιτική συνοχή. Αυτό πρέπει να είναι να, το βασικό μας μήνυμα και να επιμείνουμε σε αυτό. Και τρίτον, ήδη ε, έχουν υποθεί πολλά για τις αρχές της πολιτικής συνοχής και υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία για την περίοδο 2014-2020. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να παλέψουμε για να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση με την εισαγωγή νέων αρχών. Εντάξει, να υπάρξει απλούστευση, αλλά όχι νέες αρχές και ταυτόχρονα Παράλληλα με την ακρόαση εδώ, είχαμε και άλλη ακρόαση στην ε, Επιτροπή Προπολογισμού. Και θέλω να σας το πω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Είχαμε εκπροσώπους ε, του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μας είπε ότι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τη συμφωνία επί του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μεταξύ κρατών μελών αλλά και μεταξύ Κομισιών Κοινοβουλίου Συμβουλίου είναι τα τέλη του 19 και ακόμα καλύτερα θα ήταν πριν από τον Ιούλιο του 19 που λύγει η τρέχουσα θητεία του Κοινοβουλίου. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου όμως μας είπε ότι είναι πολύ πιθανό τα κράτη-μέλη να μην καταφέρουν να συμφωνήσουν επί του ΠΔΠ και οι κανόνες για τη μελλοντική και για να συμφωνήσουν και για του ε, μελλοντικού κανόνες της ε, πολιτικής συνοχής και ότι να περιμένουμε χρονοδιάγραμμα μόνο την άνοιξη του 20. Θα έχουμε λοιπόν την πρόταση τον Μάιο του 2018, αλλά η συμφωνία θα επιτευχθεί την άνοιξη του 2020. Και είναι πολύ αργά για να έχουμε μια ομαλή υλοποίηση ε, της πολιτικής συνοχής για την επόμενη περίοδο. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εσείς τα κράτη-μέλη σας να εργάζεστε από κοινού με τους Υπουργούς Οικονομικών και τους Υπουργούς Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης και να ε, τους συζητήσετε να πιέσουν για να έχουμε έτοιμους κανόνες και κανονιστικά πλαίσια του σημαντικών δυνατών. Το χρειαζόμαστε το 2019, όχι αργότερα, γιατί μετά και πάλι θα έχουμε καθυστερήσεις στην ε, υλοποίηση της πολιτικής συνοχής, όπως είχαμε και σε αυτήν την περίοδο. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν είδαμε έναν από τους συναδέλφους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κακώς θεωρήσατε ότι οι πλημμύρες καταστροφικές στη Δυτική Αττική δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα της πολιτικής συνοχής που συζητάμε. Η πολιτική συνοχής έχει σχέση με τις πλημμύρες και βεβαίως καθρέφτης της πολιτικής συνοχής είναι τέτοιου είδους καταστροφές. Και αν δεν γνωρίζετε τις περιοχές αυτές Μάνδρα, Μαγούλα, Νέα Πέραμο, οι 21 νεκροί και οι χιλιάδες που είναι μες στις λάσπες και προσπαθούν να περισσώσουν το βιός τους, σας υποχρέωσαν να τις μάθετε. Τι έγινε λοιπόν στη Μάνδρα και στις άλλες περιοχές και παντού με την πολιτική συνοχή. Για δεκαετίες οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι παίρναν τα κονδύλια με fast track, με επιδοτήσεις, με προνόμια, με διαδικασίες γρήγορες. Αυτή ήταν η καπιταλιστική ανάκαμψη και η καπιταλιστική ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια και την ίδια ώρα τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι εργατογειτονιές εκεί, για πολλές δεκαετίες δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν αντιπλημμυρικά έργα και μιλάμε για τους εργαζόμενους που δούλευαν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πολιτική συνοχή, γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί δεν είναι υψηλά, ε, ε, υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως το λέτε, ούτε είναι ανταποδοτικά μετά το τέλος και την ολοκληρώσή τους. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καθρέφτη είναι και αυτέ. Και βέβαια δεν έγινε μόνο στη Δυτική Αττική και σε άλλε περιοχέ έχει πλημμύρε και στην Ελλάδα και σε άλλε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε λίγο και λιγάκι. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι αυτή είναι η ανάπτυξη και το κρίσιμο ερώτημα είναι ανάπτυξη για ποιον. Για τους μεγάλους επιχειρηματικούς όμιλους που ξεκοκαλίζουν όλα αυτά τα κονδύλια που περιγράφεται όλο αυτό το διάστημα ή για το λαό. Αυτή είναι λοιπόν η, η, μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι το παραμύθι της ανάπτυξης ότι θα μοιραστεί και κάποιο ε, ψίχουλο για τους ε, εργαζόμενους και ζητάμε εδώ και τώρα αποζημιώσεις ε, και από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει μεγάλους περιορισμούς και όρια που η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει καθέσει ψήφισμα ειδικό για να αρθούν αυτοί οι απαράδεκτοι όροι και, οι περιορισμοί και να δοθούν αποζημιώσεις στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που δεν παίρνουν φράγκο όλα αυτά τα χρόνια από το λεγόμενο Ταμείο Αλληλεγγύης και ταυτόχρονα να παλέψουν οι εργαζόμενοι γιατί τίποτα δεν θα τους χαριστεί να παλέψουν για τη δικιά τους εξουσία και οικονομία που θα λειτουργεί με τις δικές τους ανάγκες και τα κριτήρια και όχι με τα κριτήρια του κεφαλαίου. Thank you. And... Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει, έχουν οι ομιλητέ μας για τα καταληκτικά του σχόλια. Ξεκινούμε από τον κύριο Αμπ. Δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσει στις θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εσά, Δεν ξέρω αν έχετε κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Πράγματι, πρέπει ήδη στις 6 να είμαι στο αεροδρόμιο. Τέλος πάντων, πρέπει να φύγω πιο νωρίς από ό,τι είχα προβλέψει. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη σημερινή ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Άκουσα ορισμένες ε, παρεμβάσεις με τις οποίες συμφωνώ απολύτως. Όλοι θέλουμε να απλουστεύσουμε τα κριτήρια χρηματοδότησης, τους κανόνες. Κανείς ε, δεν αντιτίθεται σε αυτό. Υπάρχουν όμως και απόψεις ε, που με βρίσκουν αντίθετο. Το Συμβούλιο είναι ο χώρος όπου τα κάθε μελη μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και μετά μπορούμε να τις ε, επεξεργαστούμε από κοινού και η Κομισιόν να υποβάλει νέα πρόταση. Η Προεδρία δεν, ε, δεν ισχύει μάλλον ότι η Προεδρία δεν θέλει να συνεχίσει τη συζήτηση. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε ε, να δώσουμε τη σκητάλη και στην επόμενη Προεδρία και να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τον κανονισμό Omnibus και ελπίζουμε σύντομα να επιτευχθεί συμφωνία και να σημειωθεί πρόοδος. Γιατί χρειαζόμαστε την πολιτική συνοχή. Τη θεωρούμε σημαντική Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έργο μας και να αντανακλάτε και στις αποφάσεις που θα πάρουμε και την επόμενη άνοιξη και στο μέλλον. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή πτήση. Ο κύριος Σνάιντερ, δεν ξέρω αν θέλετε να δευτερολογήσετε. Ευχαριστώ. Ε, να δευτερολογήσω. Πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ήταν κάτι που ακούστηκε πολλές φορές ε, στη συζήτηση. Εμείς θέλουμε ε, να έχουμε ένα μέρος των κονδυλίων συνοχής αναλογικά και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό ως αίτημα. Αλλά αν δεν υπάρχει ένα κονδύλι για τις πολιτικές συνοχής, ε, στο πολιετές ε, δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε για την πολιτική συνοχή. Αυτό είναι σαφές. Δεν είναι όμως αρμόδιος ο Επίτροπος Έτιγκερ για αυτά τα θέματα που έρχεται σε σας αύριο ε, και δεν είναι πρώτη φορά φαντάζομαι που έρχεται, έχει ξανάρθει και σε εμά πολλές φορές ήρθε στην Επιτροπή των Περιφερειών και είπε ότι καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ε, το θέμα μας ε, και γιατί ήταν και αυτός περιφερειάρχης αλλά δεν είναι απόλυτα αρμόδιος. Επίσης σε ό,τι αφορά τις ε, ε, περιφέρειες ε, και την επιλεξιμότητα με βάση το ΑΕΠ. Φυσικά υπάρχουν αυτά τα κριτήρια, αν μια περιοχή είναι μεταβατική, αν είναι επανάπτυκτη ή ανεπτυγμένη. Σίγουρα όμως υπάρχουν νέες προκλήσεις και υπάρχουν νέες απαιτήσει και στο πλαίσιο της ε, ε, πολιτικής συνοχής και αυτά τα προβλήματα αποδυναμώνουν ε, τη συνοχή. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη και στην πολιτική συνοχή για να μπορεί περισσότερο και καλύτερα να παρεμβαίνει στο μέλλον σε σχέση με το τι συμβαίνει σήμερα. Μεταξύ αυτών των προβλημάτων είναι τα δημογραφικά προβλήματα. Πράγματι υπάρχουν κάποιες περιφέρειες οι οποίες θα μείνουν ακόμη πιο πίσω. Τώρα για τις αρεσιμότητες. Σας είπα και εγώ ότι δεν είμαστε υπέρ. Ε, βέβαια, ε, έχουμε και την εκ ε, των προτέρων αιρεσιμότητα. Δεν ισχύει για αυτήν, γιατί νομίζουμε ότι εξάντα αιρεσιμότητα, εκ των προτέρων αιρεσιμότητα μπορεί να γίνει ένα καλό εργαλείο που να έχει θετικές το θετικό αντίκτυπο. για τον κύριο Χέτμαν, για τη δύναμη των περιφερειών, πράγματι, αυτό πρέπει να το πούμε κυρίως στα κράτη-μέλη θα, καλά θα κάνουν τα κράτη-μέλη να θεωρούν τις περιφέρειες όχι σαν ε, κάτι ενοχλητικό ε, που άντε πώς θα τους συμπεριφερθούμε κτλ. Αλλά η δύναμη τους είναι δύναμη και του κράτους. Και όσο πιο δυνατή είναι η περιφέρεια, τόσο πιο δυνατό είναι το κράτος συνολικά Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες, να μην τις ρίχνουν στον άλλον. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Εμείς ε, που είμαστε στις περιφέρειες ε, βλέπουμε ποια θεωρούμε ότι είναι καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας λέτε μας ότι και εμείς κάνουμε τα πράγματα πιο πολύπλοκα. Εμείς μιλάμε για απλούστευση. Κύριε Τσέλερ, πράγματι ε, όλοι, ε, όλα τα επίπεδα πρέπει να προχωρήσουν στην απλούστευση αυτή. Θέλω να τονίσω όμως ότι ε, έχουμε μία αλληλουχία από πάνω προς τα κάτω. Έχετε 2.000 προδιαγραφές, είπατε τώρα, ε, για τους διαχειριστικούς φορείς. Ε, αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν στο τοπικό επίπεδο. Υπάρχει όμως και ο έλεγχος. Και εκεί έχει βγει εκτός έλεγχου η κατάσταση. Ε, μπορεί κανείς ε, με αυτό τον υπερβολικό έλεγχο τελικά να επιβαρυνθεί τόσο πολύ που ε, επειδή οι διαχειριστικές αρχές λόγω του μεγάλου ελέγχου φοβούνται μην κάνουν κάποιο λάθος δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και στις εθνικές ελεγκτικές αρχές βέβαια. Και εμείς ίσως θα μπορούσαμε έτσι να βοηθήσουμε την απλούστηση. Και το τελευταίο και εμείς, ε, το έχω πει και εγώ, μιλάμε για τα προβλήματα, για τις αδυναμίες και για τα αρνητικά που σχετίζονται με την πολιτική συνοχή. Θα ήθελα όμως στο τέλος να τονίσω ότι τα διαφορετικά ταμεία, η πολιτική συνοχή είναι μια ιστορική επιτυχία, τεράστια επιτυχία στην ανθρώπινη ιστορία. Ποτέ δεν υπήρξε κάτι σαν ε, την πολιτική ε, συνοχή που να είναι ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο αλληλεγγύη. Πρέπει να είμαστε λοιπόν υπερήφανοι και με μεγάλη περηφάνεια να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε αυτό το εργαλείο και ελπίζω ότι η Βουλγαρία που θα έχει την Προεδρία ε, να φέρει τη δάδα της πολιτικής συνοχής ψηλά. Thank you. Thank you Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σνάιντερ, Ευχαριστούμε για τον εξαιρετικό αυτό λόγο και ελπίζω πραγματικά να συνεχίσουμε μαζί γιατί όπως αναφέρει η Βουλγαρική Επερχόμενη Προεδρία ισχύει εν Κυρία Πλούμ θέλετε να επανέλθετε. Ναι βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ρουμανικά. Συμπερασματικά λοιπόν, μετά τη σημερινή συζήτηση που ήταν πολύ θετική, όλοι όσοι πήραν τον λόγο, όλοι εμείς λοιπόν είμαστε υπέρμαχοι της πολιτικής συνοχής και θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ένας από τους ε, πυλώνες της επενδυτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό χάρη στην προστιθέμενη αξία, την οποία αποδεικνύει ξανά και ξανά. Προφανώς και χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και προβολή των αποτελεσμάτων ε, της ε, πολιτικής συνοχής σε ό,τι αφορά ε, τις ωφέλειες που εξασφαλίζουμε έτσι για την καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Σημείωσα επίσης ότι όλοι θεωρούμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην ε, υλοποίηση της ε, πολιτικής συνοχής. Αυτό είχα επισημάνει και στην αρχική μου παρέμβαση. Εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών, των δικαιούχων, σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε μαζί να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα και κάθε φορά αυτό αποδεικνύουμε. Δείχνουμε λοιπόν ότι με την ένωσή μας, με τις κοινέ προσπάθειες όλων των Ευρωπαίων, καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. Και κάθε φορά η απάντηση ε, που δίνουμε στις προκλήσεις εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουμε μέτρα. Όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι μαζί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μαζί με τους Ευρωπαίους πολίτες, με την Επιτροπή των Περιφερειών. Πιστεύω ότι ε, πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την πολιτική συνοχή στην οποία χρειαζόμαστε όλοι. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω ε, την κυρία Κρέλ για τον τρόπο με τον οποίο κάθε φορά υπογραμμίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι και οι πραγματικοί κερδισμένοι από την ε, πολιτική συνοχή και την περιφερειακή μας πολιτική. Πολύ χρήσιμη αυτή η παρατήρηση. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα με τον άλλον, να υπάρχει καλύτερο συντονισμό και αυτό απευθύνεται και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνεργασία μεταξύ ημών για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κωσίλεβα έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Μιχαήλοβα. Με εντυπωσίασαν και εμένα τα όσα είπε ο κύριος Σνάιντερ για την επερχόμενη προεδρία μας. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα αυτό. Μας εμπνέει όλους ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, τη συνεργασία, τις συνομιλίες. Να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Η Βουλγαρία είναι ένα πολύ καλό μέρος για τέτοιες συζητήσεις, διότι όπως είπα είμαστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά χρήσιμη, ορατή πολιτική που αρέσει στον κόσμο. Όλοι συμφωνούν ότι έχει συμβάλει στη βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης στη χώρα μου. Έχει βελτιώσει τις μακροοικονομικές συνθήκες και την οικονομία της χώρας. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο εμείς ε, οι άνθρωποι, περισσότεροι από εμά να διαδίδουμε αυτό το μήνυμα. Να εξηγούμε στον κόσμο τι είναι η πολιτική συνοχής. Τι συμπεραίνω από τις συζητήσει που άκουσα σήμερα το απόγευμα και ευχαριστώ που μου δώσετε και αυτή την ευκαιρία να συμμετέχω. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για μένα. Τι συμπεραίνω λοιπόν πρώτα απ' όλα όλοι συμφωνούμε ομόφωνα ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να συνεχιστεί. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει το στοιχείο της πολιτικής συνοχής. Ναι, γιατί τα χρηματοδοτικά μέσα να υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παντού. Πρέπει να υπάρχει επίσης ευελιξία και απλούστευση. Η απλούστευση θα πρέπει να βελτιωθεί φυσικά, να αναβαθμιστεί, διότι ήδη σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι το σημαντικότερο κομμάτι του κανονισμού. Η ευελιξία θα πρέπει να καταλάβει πιο σημαντική θέση στο επερχόμενο πακέτο. Η ευελιξία σε όλες τις πτυχές, διαδικασίες, κανόνες, συνδυασμοί, δυνατοί, όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότητα, σε αποτελέσματα. Και θέλω και πάλι να τονίσω το, το χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος. Πρέπει να δράμε έγκαιρα, ανταγωνιστικά ισχυρά ενωμένα. Αλλά ενωμένα, αλλά πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί, οπότε τα πράγματα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ξανά όλους σας. Ελπίζω να σας δω σύντομα στη Βουλγαρία για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες Έχουμε συναντήσει ε, στη Βουλγαρία στις αρχές του επόμενου χρόνου και διαφορά φόρουμ για την πολιτική συνοχή. στο πλαίσιο της επερχόμενης πρότασης της Κομισιόν για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Περιμένω με ανυπομονησία να συνεχίσουμε με τόσο θετικό πνεύμα τις συζητήσεις αυτές και να έχουμε και την ευκαιρία να αρχίσουμε να εργαζόμαστε μέσα στην επόμενη προγραμματική περίοδο από την πρώτη της ημέρα. Ευχαριστώ και ξανά και πάλι όλους σας. Ήταν μεγάλη μου χαρά που βρέθηκα εδώ μετα... ανάμεσά σας. Ευχαριστούμε. Κυρία Κρέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Μια παρατήρηση καταληκτικά και εγώ προσβλέπω με υπομονησία την ε, Βουλγαρική Προεδρία. Ήμουν με μια αντιπροσωπεία στη Σόφια και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή δέσμευση και προσήλωση για μια καλή και αποτελεσματική πολιτική συνεχίση και αυτό είναι το σωστό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από την Βουλγαρική Προεδρία. Επίσης ε, χαίρομαι που είναι εδώ η κυρία Πλούμπα γιατί και με ε, την αντιπροσωπεία που μάλλον και, και στη Ρουμανία πήγαμε μια αντιπροσωπεία και νομίζω ότι βλέπουμε στις χώρες αυτές θετικά παραδείγματα. Υπάρχουν, τα είδα με τα μάτια μου, ότι έχουμε πολύ ε, καλή, ε, καλά αποτελέσματα. Έχει επίδραση η πολιτική συνοχή επιτόπου στα κράτη. Μία παρατήρηση. Θα είδατε ε, και θα παρατηρήσατε ότι λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε προς το τι θέλουμε. Εκτός όμως των αιθουσών του Κοινοβουλίου είναι πολλοί αυτοί που δεν τα βλέπουν τα πράγματα όπως εμείς και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε αγώνα και εντός Κοινοβουλίου ε, και με τα κράτη-μέλη και με ε, την Κομισιόν και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε υποστήριξη αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η πολιτική συνοχή ε, έχει αποτέλεσμα και ρέουν τα κονδύλια. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να διατίθενται κονδύλια μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τα οποία τελικά δεν ε, χρησιμοποιούνται και γυρίζουν πίσω λίγο πολύ. Ε, πώς μπορεί κανείς έτσι να δικαιολογήσει ένα υψηλότερο προϋπολογισμό για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Δεν έχει ισχυρά επιχειρήματα, δεν μπορεί να απαιτήσει περισσότερα κονδύλια αν δεν υπάρχει αξιοποίηση των ήδη ε, διατεθέντων. Αυτά είχα να πω και προσβλέπω στην μεταξύ μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ το προνόμιο σε εσά, κύριε Φονμπρέσκα, να είστε ο τελευταίο ομιλητή για σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πιστεύω ομόφωνη υποστήριξή σας προς την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ που μας υπενθυμίζετε και πόσο σημαντική είναι για τους πολίτες, διότι βασίζεται στη συνεργασία και αφορά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Όπως ορισμένοι από σας τονίσατε, δυστυχώς αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν γίνεται πάντα γνωστή. Είναι σημαντικό λοιπόν και για μα, ε, στην Κομισιόν, σε όσου ασχολούμαστε με την πολιτική συνοχή, για να έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο σε αυτέ τις κρίσιμες εποχές όπου υποτίθεται ότι προετοιμάζουμε τον επόμενο προπολογισμό και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όπω είπα θα ε, τεθεί προς συζήτηση την Άνοιξη του 2018. Ευχαριστώ για όλη σας τη συμμετοχή, όλες τις συμμετοχές. Θα λάβουμε υπόψη τα σχόλιά σα στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Ήταν, υπήρξαν κάποιες πολύ χρήσιμες συστάσεις. Ήθελα να πω, ε, να αναφερθώ σε δύο-τρία θέματα όσον αφορά την αιρεσιμότητα. Για άλλη μια φορά το παρακάναμε. Αυτό είναι αναμφίβολο. Πρέπει όντω να μειώσουμε σαφώ την αιρεσιμότητα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι για ορισμένα ζητήματα, για ορισμένε επενδύσει, πώς να τις πω, δράσεις προτεραιότητας είναι απαραίτητες κάποιες προϋποθέσεις. Ε, για παράδειγμα, στη μεταφορά εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε με πολλά χρήματα τις μεταφορές σε πολλά κράτη-μέλη και ανακαλύψαμε ότι σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν κεντρικά σχέδια για τις μεταφορές. Πώς γίνεται να επενδύουμε δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα των μεταφορών χωρίς να γνωρίζουμε ποια είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της χώρας αυτής για τις μεταφορές. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι αυτές οι οποίες θέλουμε να εστιαστούμε στο μέλλον. Ένα δεύτερο ζήτημα η απλούστευση. Δεν πρόκειται να κάνουμε επανάσταση, αυτό είναι σαφές. Μια απλή εξέλιξη όμως δεν θα ήταν ε, επίσης επαρκής. Η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι ότι ε, μελετάμε τον κανονισμό άρθρο προς άρθρο και αναρωτιόμαστε, χρειαζόμαστε αυτό το άρθρο, διότι ορισμένα από αυτά τα έρθρα πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι σας ε, όσοι έχετε ασχοληθεί με προγράμματα ξέρετε ότι τα προγράμματα μπορούν να δαπανίσουν λεφτά μόνο στο προγραμματικό, στην, στην περιοχή του προγράμματος. Δηλαδή αν είναι στο Βραδεμβούργο, μόνο στο Βραδεμβούργο. Αλλά σε τελική ανάλυση αυτό δυσκολεύει τα πράγματα, τα κάνει πιο περιπλόκα. Ναι, υπάρχουν και ορισμένε εξαιρέσει. Δεν μπορεί κανεί. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τον προπόστο να μην ξοδεύει κανεί τα χρήματα εκτό τη περιφέρεια. Αλλά αν οι εταίροι του προγράμματο συμφωνούν ότι θέλουν να ξοδέψουν ε, τα χρήματα για μια ας πούμε ε, εμπορική έκθεση στην Κίνα για να προβληθούν, ε, για να αυξήσουν τη δουλειά τους. Για ποιο λόγο εμείς να το αμφισβητήσουμε. Εφόσον οι εταίροι του προγράμματο του συμφωνήσουν, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν τέτοιοι κανόνε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι παρά ένα παράδειγμα. Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό στην άνοιξη του 2018 και ελπίζουμε να σας πείσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τους ελέγχους και τους οικονομικούς ελέγχους. Σε έναν τέλειο κόσμο τι θα κάναμε θα βασιζόμασταν στους εθνικού κανόνε, διότι οι εθνικοί κανόνε είναι αυτοί που γνωρίζουν οι εθνικές διοικήσεις και οι δικαιούχοι, και οι δικαιούχοι γιατί για τις περισσότερες δαπάνες οι οποίες είναι εθνικής φύσης δεν μπορείτε να έχετε από τη μια το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη το εθνικό εγχειρίδιο και να ψάχνετε να βρείτε ποιοι κανόνες ισχύουν. Δεδομένου αυτού είναι επίσης σαφές ότι δεν μπορούμε, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε μια κατάσταση όπου δεν γνωρίζουμε πλέον καθόλου τι συμβαίνει με τα χρήματα αυτά, γιατί όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό σε τελική ανάλυση και πρέπει να έχουμε κάποια διασφάλιση ότι ό,τι συμβαίνει στις περιφέρειες και σε τοπικό επίπεδο τηρεί κάποια πρότυπα. Τι σημαίνει αυτό, ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά όπως είπα, στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε στις περιπτώσεις όπου αντιλαμβανόμαστε ότι οι διοικήσεις, οι τοπικές και οι περιφερειακές καταλαβαίνουν να χειριστούν τα κονδύλια, καταφέρουν να χειριστούν τα κονδύλια χωρίς επίβλεψη από τις Βρυξέλλες, τότε θα πρέπει να τους δείξουμε εμπιστοσύνη. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να ρυθμίσει κανείς με νόμο την εμπιστοσύνη. Μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, αλλά δεν μπορεί να την νομοθετήσει. Ε, άλλα δύο πράγματα, συγγνώμη που μακρηγόρησα τώρα, για τα κριτήρια κατανομής. Πρέπει να τους ρίξουμε μία ματιά. Ε, πολύ επικριτική. Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στο ΑΕΠ ως κριτήριο μόνο. Θα είναι σημαντικό κριτήριο ανεξαρτήτως, αλλά πρέπει να δούμε και τις νέες προκλήσεις και να δούμε σε ποιο βαθμό η πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Είτε μιλάμε για κοινωνική ένταξη, είτε για κοινοτομία είτε για ενέργεια και κλίμα και όλα αυτά. Και τέλος, η ευελιξία και η εστίαση στο αποτέλεσμα. Άκουσα πολλούς από εσά να διαμαρτύρεστε για, την, για το ανέλικτο της πολιτικής αυτής. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε κάποιες ριζοσπαστικές ιδέες, ότι για παράδειγμα στο μέλλον ε, να προγραμματίσουμε μόνο τα τέσσερα πρώτα χρόνια του επτά δημοσιονομικού πλησίου και μετά να πούμε θα γίνει μια αναθεώρηση μετά από αυτή την περίοδο και μετά θα δούμε μαζί κατά πόσο χρειάζεται για παράδειγμα να ανταμείψουμε, να βραβεύσουμε αυτούς που έδειξαν καλές επιδόσεις αν υπάρχουν νέε προτεραιότητε. Σκεφτείτε τι έγινε με τη μετανάστευση. Προτεραιότητε τι οποίε δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο κατανομή των κονδυλίων και δαπάνη του. Ε, αυτό όμω θα είναι μια έκπληξη που σα επιφυλάσσουμε για του χρόνο Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να περιμένουμε ορισμένε εκπλήξεις για την επόμενη χρονιά. Ελπίζω όχι πάρα πολλέ. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη συμμετοχή τους σήμερα στη συνεδρίαση. Σας διαβεβαιώ ότι εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, τις εμπειρίες σας, τις θέσεις σας, τη στήριξή σας προς ε, το έργο μας για την πολιτική συνοχή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, τη σημερινή συνάντηση. Ελπίζουμε να μείνουμε σε επαφή. Ακούσαμε πολλές ε, γνώμες και απόψεις από εθνικές κυβερνήσεις και κοινοβούλια και σας ευχαριστώ. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα αναζητούμε το καλύτερο δυνατό μέλλον για την πολιτική συνοχή. Θέλουμε να βρούμε μια απλή, αποτελεσματική πολιτική συνοχή με γνώμονα τα συμφέροντα και τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, πιο ανοιχτή, πιο ευέλικτη, πιο κατανοητή. Μια πολιτική που θα επενδύσει στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ενωμένοι Μπορούμε να, να το πετύχουμε αυτό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ε, έχουμε πολύ καλή εμπειρία ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, πρόταση Omnibus. Γιατί δεν παρουσιάζεται και εκεί επαναστατικέ ιδέε. Ξέρω ότι η Επιτροπή είναι πολύ αυστηρή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αστειεύομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σα. Πολύ γόνιμος ο διάλογο σήμερα. Ελπίζω να επαναληφθεί και με μεγάλη χαρά να σα υποδεχθούμε εκ νέου στο μέλλον στο Κοινοβούλιο. Η Πρόεδρο ευγενικά ευχαριστεί και τους διερμηνεί. εμείς. Μας βοήθησε, να να επικοινωνήσουμε και να νιώσουμε όλοι πιο άνετα τη μετρική μας. Πέρα συνεδρία σας. Καλό σας βράδυ.